Euh, Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους μας από το Νότιο Σουδάν οι οποίοι μας έδωσαν τη χαρά να έρθουν να παραστούν σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Με κάθε, ε, λοιπόν, πάρα πολύ ειλικρινά, σας εύχομαι καλώς ήρθατε. Nous allons notre ordre jour. Λοιπόν, έχετε σχόλια για αντιρρήσεις προς το σχέδιο της μερισιάς διάταξης. Όχι, επομένως εγκρίνεται. Έχετε λάβει τα πρακτικά συνεδρίασης της 21ης-22ης Ιανουάριου 2013. Αν έχετε παρατηρήσεις ε, ότι αυτά τα πρακτικά, σας παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά τη γραμματεία μέχρι τη σημερινή, το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Αν δεν έχετε σχόλια θα εγκριθούν τα πρακτικά ως έχουν. Les recommandations émises et les décisions prises Έχετε στο φάγγελό σας τις συστάσεις ε, και τις αποφάσεις από τη συνεδρία των συντονιστών, τη συνεδρία των συντονιστών της 19 Φεβρουαρίου. Αν έχετε παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα, μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά την γραμματεία πριν το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, αλλιώς θα εγκριθούν ως έχουν τα αποτελέσματα της συνεδρίας των συντονιστών. Έχω δύο ανακοινώσεις. και θα εκμεταλλευτώ το χρόνο που έχω ε, στη διάθεσή μου για να αναφερθώ στο ζήτημα του AIDS. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο στις αναψώμενες χώρες σε ό,τι αφορά την ανείχνευση. Όμως ε, η Ποσαχάριος Αφρική Έχει πολύ βελτιωθεί, αλλά έχουμε 14,1 εκατομμύρια παιδιά θύματα, ε, μάλλον έχουν χάσει έναν ή δύο γονείς ε, λόγω του HIV και του AIDS. Επειδή βλέπουμε ιδίως στη Βόρεια Αφρική ε, να οξύνεται η επιδημία αυτή. Όμως η καταπολέμηση του HIV-AIDS θα πρέπει να είναι μια πολιτική την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και να συμπεριλάβουμε σε όλους τους τομείς της αναπτυξική μας πολιτικής. Είναι μια πολιτική για την, ε, που πεντάστες στην επιτεκτό στόχο τη χιλιετίας. Υπάρχει όμως ε, ανησυχία και αβεβαιότητα και ω προς τα ποσά αναθεματική ε, και συνεχίζονται και συζητήσει για τον προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε ώστε τουλάχιστον να το 20% του ΦΕΤ και του ειδικού αναπτυξιακού μέσου DCI να αποδοθούν ε, για την βασική εκπαίδευση και θέλουμε επίσης ένα σημαντικό ποσό των εσόδων από το μελλοντικό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να πηγαίνουν στην ανάπτυξη και ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη. Γνωρίζω ότι αγαπητοί συνάδελφοι όλοι σας είστε ευαισθητοποιημένοι στα θέματα αυτά Ξέρω ότι οργανώνεται συχνά εκδηλώσεις ε, για αυτό το θέμα και για το έτσι, ιδιαίτερα και για τις άλλες μοδοτικές γνώσεις και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά τη σημασία την οποία αποδίδουμε στην τραγωδία αυτή. Και ιδίω λαμβάνοντα υπόψη ότι παρά τι δεσμεύσει που έχουν ληφθεί, το σχετικό ε, μέρο ε, του προπολογισμού το και το 2010 έχουν πέσει κατά 8,2 ε, μάλλον από το 8,2 στο 7 το 2010 τα αποδεδόμενα ποσά. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος ανακοίνωσης και για το δεύτερο σκέλος θα ήθελα εν συντομία να σας μιλήσω για το Αφγανιστάν και τη διαφθορά στο Αφγανιστάν. Την Τρίτη, το ειδικό δικαστήριο που έχει συγκροτηθεί στην Καμπούλ για την υπόθεση της Καμπούλ Μπάνκ, όπου 900 εκατομμύρια τα οποία είχαν δοθεί από τα δημόσια αφαιρέθηκαν είχαν δηλαδή στηρίξει αυτά τα χρήματα τα οποία προέρχονταν στο μεγαλύτερό τους μέρος από τη διεθνή κοινότητα από εμάς είχαν αφαιρεθεί για να στηρίξουν την τράπεζα. Τώρα έχουμε την ε, αυτή ε, για την υπόθεση υπήρξε απόφαση για νοθεία και πλαστογραφία ε, εγγράφων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ε, καταδικάστηκαν από το ειδικό αυτό δικαστήριο οι ένοχοι, αλλά μόνο για κατάχρηση εμπιστοσύνη και όχι για ε, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πέντε αιτής κάθερξη ήταν το αποτέλεσμα. Τα μισά χρόνια ήταν σε πολυτελή ξενοδοχεία προσωρινή κράτηση. Δεν υπήρξαν κατασχέσεις περιουσιών, δημεύσεις ε, περιουσίας. Εγώ έκανα λόμπι να υπάρξει έφεση στην απόφαση αυτή, διότι διακυβεύονται πολλά. Γιατί αυτή, με αυτή την καταδίκη ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, το μηχανισμός ο οποίος ισχύει για το ξέπλυμα χρήματος. Και επίσης με ενοχλεί και ιδιαίτερα το θέμα που, της μη δίμευσης, πώς μπορούν να ε, επιστραφούν αυτά τα ποσά ή να καλυφθούν με άλλο τρόπο. Μήπως ακριβώς αυτό ήταν ο στόχος τελικά. Υπάρχει έφεση, η έφεση βλήθηκε απόφαση. Είναι σημαντικό αυτό για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας μεγάλος χρηματοδότης και δωρητής και δεν θα ήθελα εγώ να εξαφανιστούν ε, σε συγκεκριμένες τσέπες αυτά τα 900 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Σταματώ εδώ και είναι το λόγο στον κύριο Γκέρενς. Κοιτάξτε. Ποιος? Ο Καρζά είναι αναμειγμένος στην όλη υπόθεση. 30 εκατομμύρια δολάρια δάνεια πήρε που δεν είχε πρόθεση να επιστρέψει. Ο αντιπρόεδρος και αυτός ενεπλάκη είναι η πρώτη φουρνιά αποφάσεων αυτή που ελήφθη και οι μισθωτοί της ε, τράπεζας, οι διευθυντές της τράπεζας και οι επικεφαλής των ελεκτρικών αρχών ήταν αμειγμένοι. Ο Γενικός Αγγελέας παρετήθηκε μετά τις ε, αποφάσεις. Υποσχέθηκε ότι δικαιούχε οι μέτοχοι των τραπεζών, ε, όσοι έχουν παρατυπήσει εδώ ε, των, τραπεζών και οι μέτοχοι θα διωχθούν. Και αυτό θα το παρακολουθήσει η διεθνής κοινότητα από κοντά, το πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Κυρία Ντεκάιζερ, ευχαριστώ κυρία Προέδρε για τις πληροφορίες, τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν είμαι νομικός. Αναφερθήκατε σε ειδικό δικαστήριο αυτή τη φορά. Η προσφυγή σε ποιο δικαστήριο γίνεται. Απάντηση. Το Αφγανιστάν δημιούργησε ειδικό δικαστήριο για να επιληφθεί το θέμα τους. Δε 900 εκατομμύρια δολάρια είναι τεράστιο ποσό. Πρωτοφανές. Και μάλιστα και σαν ποσοστό του εσωτερικού καθαρίστου προϊόντος. Υπήρχαν πολλά κενά στη θεσπιστή νομοθεσία. Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν θα πήγαινε στο εφετείο, τι είδου θα ήταν η προσφυγή που θα μπορούσε να γίνει. Ο πρόεδρος του εφετείου είπε ότι υπάρχουν δύο επίπεδα, το κανονικό εφετείο, δικαιοδοτικά, και μετά το ανώτατο δικαστήριο. Τώρα έχει δρομολογηθεί η έφεση. Ας ελπίσουμε ότι δικαστικό σύστημα θα μπορέσει να εφαρμόσει καλύτερα ε, την νομοθεσία από ό,τι έκανε στην φάση την πρωτόδικη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια σχόλια. Λοιπόν, να δώσω το λόγο. Και κλείνει το μικρόφωνο της Πρόεδρου και δεν ξέρω σε ποιον δίνει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να σας πω ότι θετήσαμε ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά τη βελτίωση της διατροφής στον κόσμο. Η ανακοίνωση έχει τίτλο «Βελτίωση ε, της διατροφής των παιδιών και γενικά διατροφής στο, στο πλαίσιο εξωτερικής βοήθειας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση». Δεν θέλουμε να να υπάρχουν φαινόμενα που δεν αναπτύσσονται σωστά τα παιδιά, να αποφεύγονται αυτά τα φαινόμενα και να μην είναι και καχεκτικά τα παιδιά, να αναπτύσσονται κανονικά με άλλα λόγια. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη θέση σωστή διατροφή. Δράση επίπεδο γλωσσών. Θέλουμε να βελτιώσουμε και τεχνογνωσία στον τομέα. Βασικά στοιχεία τη ανακοινώσεω. Θα παρακολουθούμε πολυτεμιακή προσέγγιση. Θα ακολουθήσουμε. Ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση θα αλληλοσυνοδεύονται. Από εκείνο ετοιμάσαμε την ανακοίνωση στου γενικού διευθυντέ που είναι υπεύθυνοι για την άπτυξη ανθρωπιστική βοήθεια και θα καλέσουμε τι κυβερνήσει να επιληφθούν των ευθυνών του και να ασχοληθούν με του πληθυσμού του. Και να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε πολιτικά στα πλαίσια γενικότερη προσπαθία να υποστηρίξει τι χώρε εταίρου να μειώσουν τον αριθμό των παιδιών κάτω από 5 ετών που υποφέρουν από κακή ανάπτυξη. Και 10% από τα 7 εκατομμύρια παιδιά Θέλουμε λιγότερα παιδιά μέχρι το 2025 να υποφέρουν αυτά τα φαινόμενα της μίσος της ανάπτυξης και το να μην είναι καχεκτικά. Αυτό έχω να πει για την ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μαρτίνες, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακοίνωση αυτή, η οποία αντιστοιχεί με σημείο 4 τη διάταξης. Αλλά δεν ξέρω, μήπως δεν κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω ότι όταν εσείς του δώσατε το λόγο, του το δώσατε για να ακούσετε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το προηγούμενο θέμα. Δηλαδή, σε σχέση με αυτά τα οποία μας είπατε εσείς. Μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση μας κάνατε, συγκεκριμένα για αυτή τη δίκη στο Αφγανιστάν. Μίλησε ο κύριος Γκέρνης από αυτού και νόμιζα, ε, ναι και η κυρία Ντεκάιζερ, εγώ δεν έλαβα το λόγο βέβαια, αλλά νόμιζα ότι όταν απευθυνθήκατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει την άποψή της, νόμιζα ότι ήταν γι' αυτό, γι' αυτό το θέμα. Και όχι ότι θα πρόκειται για μια διαφορετική ανακοίνωση, δηλαδή ότι θα είχαμε περάσει ήδη στο σημείο 4 τη Μέρσια διάταξη. Ναι, καλό και ενδιαφέρον και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν η Κομισιόν έχει να μα πει κάτι, ναι ή όχι, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που μα επισημάνατε εσεί με τη δική σα ανακοίνωση, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, επειδή είχα αυτό το λεπτό, αν θέλετε, για τι ανακοινώσει του Πρόεδρου, εποφελήθηκα για να πω αυτά που είπα, αλλά αυτό είναι ένα πραγματικά άλλο σημείο τη μερικής διάταξη. Ε, και στο πλαίσιο αυτού του σημείου, διά, ε, του σημείου της μερικής διάταξης μας έκανε αυτή τη σημαντική ανακοίνωση ο πρόσωπος της Κομισιόν, τον οποίο και ευχαριστώ. Τώρα, Περνάω σε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσει, δεν υπάρχουν. Οπότε θα περάσουμε στο σημείο 7 τη ημερησία διάταξη που είναι η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο γνωμοδότηση, το οποίο θα συντάξουμε για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Σαρλ Γκέρεν είναι συγητή, είναι ο συντάκτη γνωμοδότηση και θα του δώσω ευθύ αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για γνωμοδότηση. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι η καθήλυνα αρμόδια. Βλέποντας τι τελευταίες στατιστικές από το 2011 δηλαδή είχαμε πάνω από 12.000 θέσει ασύλου σε 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από παιδιά κάτω των 18 που φτάνουν μόνα τους ε, στην Ευρώπη ή τέλο πάντων φτάνοντας ε, καταλήγουν μόνα τους. Πολλές φορές αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, οργανωμένου εγκλήματος ή σωματεμπορίας. Ε, έτσι λοιπόν ε, οξέ, με οξύ το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά όλα τα κράτη-μέλη τους προτείνεται υποδοχή και, και μέρημνα, αλλά είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη που έχουν όμως προσυπογράψει τη Σύμβαση των Αμερικανών για τα δικαιώματα του παιδιού, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν ε, υπογράψει το θεμελιώδη χάρτη ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν λοιπόν μέσα ε, που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους, έχουμε την οδηγία για τη σωματεμπορία, για το άσυλο κτλ. Όμως, δεν υπάρχει ένα συνολικό μηχανισμό δεσμευτικό που θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων, την προστασία του, την υποδοχή του, την μέρημνα ε, που θα πρέπει να του παρέχεται. Το 2010 ενέκρινα ένα σχέδιο δράση η Κομισιόν για του ασυνόδευτου ανηλίκου. Θα έπρεπε αυτό να καλύπτει την περίοδο από το 2010 στο 2014 και εγκρίθηκε στα πορίσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2010. Έχοντας επίγνωση του κατεπήγοντος του όλου προβλήματος για τους ανηλίκους στα συνόδευτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να επιληφθεί αυτού του θέματος και να συντάξει μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας. Κυρία ε, Λίσμπεκ είναι η συντάκτρια της έκθεσης αυτής αντιπροπορτικών ελευθεριών. Και εμείς, όπως και οι συγγύτεροι, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή τη Επιτροπής Απολικών Ελευθεριών αλλά μάλλον βλέπουμε να είναι πιο πολύ περιγραφική παρά ε, ενεργητική πρόταση. Και κάνουμε τι εξή προτάσει. Εμεί πρώτον, αν θέλουμε να τεθεί ένα τέρμα ε, στην ασυνέπεια που υπάρχει μεταξύ των 27 πολιτικών, είναι αναπόφευκτο και απαραίτητο από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται ουτοπικό, γιατί θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την, πολιτική, την κοινή πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τα ε, σχόλια των συναδέλφων, αλλά και κυρίως τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνεί η Κομισιό να έχουμε ένα πραγματικά ε, νομικό μέσο που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που άπτονται των ε, ασυνόδευτων ανηλίκων. Και το οποίο ζητά και εισηγήτρια από την Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή. Συμφωνούμε όλοι, πιστεύω, ότι απότατο στόχος όλων των μέτρων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους παραμένει να εντοπιστούν, αλλά βέβαια πάντοτε προς το συμφέρον τους, ε, λύσεις βιώσιμες. Ίσως ε, μία από αυτές θα ήταν η επιστροφή στη χώρα προέλευσής τους, ε, η εγκατάστασή τους σε μια τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων. Από τη δική μας πλευρά, την αναπτυξιακή, εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες με την προοπτική της υποδοχής και της ε, ανάληψης της ευθύνης για τους ασυνόδευτους ανηλίκων και αποτροπή ουσιαστικά της ε, εισόδου ε, των ατόμων αυτών. Θα πρέπει όλα αυτά βέβαια να τα δούμε και από το γενικότερο πρίσμα και της πολιτικής μετανάστευσης ασύλου. Και θα πρέπει στην ε, ατζέντα, στο θεματολόγιο διαλόγου που έχουμε με τους εταίρους μας, τη χώρες, περιλάβουμε αυτά τα θέματα. Και επειδή έπρεπε να καθορίζονται τα χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα του ασύλου και τη μετανάστευση αυτόν τον καιρό, θα θέλαμε να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στα ζητήματα των ασυνόδευτων ανήλικων. Η προστασία των παιδιών δυστυχώ αυτή τη στιγμή ε, εντάσσεται στην ανθρωπιστική πολιτική, ε, αλλά έχει τη λιγότερη χρηματοδότηση. Και εμείς ζητούμε να εισαχθεί ένα συντονισμένο σύστημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή δεδομένων, να ενισχυθεί και ο ρόλος της Frontex και της Europol και επίσης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης να συμμετάσχει και αυτό. Ευχαριστώ. Κύριο Βένσον, έχετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Βένσον, δεν τον ακούμε. för i mitt tycke mycket bra yttrande. Det är lätt att hålla med om allt som står i yttrandet. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ σωστά αυτά που ακούσαμε. Θα υποβάλουμε βεβαίως και εμείς τις ε, τροπολογίες μας, αλλά αυτές ε, θα βοηθήσουν για να ενισχυθεί η έκθεση και να συμπληρωθεί σε κάποια σημεία. Θέλω να πω κάτι, κυρία Πρόεδρε. Είναι όντως σημαντικό το θέμα αυτό. Τα τελευταία δέκα χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν εξαφανιστεί δεκάδες χιλιάδες παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους. 300 παιδιά εξαφανίστηκαν μόλις το 2012. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να πω και πώς να το πω. Ε, πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική σε ό,τι αφορά το άσυλο και τους πρόσφυγες. Ε, δεν μπορούμε να αφήνουμε τα παιδιά που είναι πρόσφυγες να εξαφανίζονται κάπου. Ε, πρέπει να βρεθεί μια σωστή πολιτική. Δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να, έχουμε, να δώσουμε σημασία στα νούμερα. Και επίσης άλλο ένα σημείο. Αν ε, όταν συζητούμε το θέμα αυτό, μιλούμε για ροές, ε, ε, και για κατανομή βαρών. Ε, δηλαδή τους θεωρούμε βάρος αυτούς τους ανήλικους, έτσι όπως το συζητούμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι απλώς ε, μετατρέπονται σε στατιστικά στοιχεία, σε βάρη που πρέπει να καταναμηθούν σωστά, σε, μετατρέπονται σε αριθμούς, ενώ δεν είναι. Είναι άνθρωποι. Μιλούμε για ανθρώπους. τα περισσότερα αναθεμελιώδη δικαιώματα δεν, ε, δεν μπορούμε να τα καταπατούμε, δεν μπορούμε να, να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι παράνομοι. Δεν είναι παράνομοι οι άνθρωποι ως άνθρωποι, είναι παράνομο αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να θέτουμε ένα αμφιβόλο τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Μιλούμε για ελευθερία, για ασφάλεια, Αυτά τα πράγματα δεν υποκαθίστανται από τίποτε και αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια και πάντα το λέει και η Κομισιόν στις ανακοινώσεις της. Παρόλα αυτά είμαστε πάντα πολύ μακριά από το να έχουμε επιτύχει την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την ε, χώρα τους ε, για να ε, ζώσουν τη ζωή τους, για να βρεθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και επίσης σε ό,τι αφορά την κοινωνική πτυχή της υπόθεσης ε, τα περισσότερα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους και είναι παιδιά προσφύγων στις ευρωπαϊκές χώρες, αυτά τα παιδιά δεν έχουν επιλογή. Ε, να δεν μπορούν να διαλέξουν, δεν έχουν άλλη λύση για να ζήσουν. Οπότε είτε θα πεθάνουν είτε θα φύγουν από τη χώρα τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σωστή πολιτική ε, για τους πρόσφυγες, για το άσυλο, μια σωστή πολιτική η οποία δεν θα έχει ως μόνο στόχο να στείλει αυτούς τους ανθρώπους πίσω το, το γρηγορότερο δυνατόν ή του, τα παιδιά αυτά να τα στείλει πίσω σε εμπόλεμες ζώνες. Μία πολιτική για την ε, ε, μετανάστευση θα πρέπει να δει τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θεωρούνται ως άνθρωποι που έχουν αξιοπρέπεια δεν μπορούμε να τους περιγράφουμε και να τους θεωρούμε ως βάρος. Είναι άνθρωποι που έχουν ελπίδες, που έχουν όνειρα, που έχουν οράματα. Κάθε πρόσφυγας είναι ένας άνθρωπος και αυτό είναι δική μας ευθύνη να το εδραιώσουμε. Πρέπει να τους προσφέρουμε ασφάλεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν μια σωστή πολιτική. Και αυτό ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο έχει ζήσει κάποιος σε μια χώρα. Όπως είπα θα υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες ε, στο κείμενο του κυρίου Γκιόρενς σε ό,τι αφορά τα θέματα της μετανάστευσης, αλλά θεωρώ ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο να τον καλύτερα τα εργαλεία που έχουμε ήδη στα χέρια μας πριν θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απλά ένα βάρος. Πρέπει να τους θεωρούμε ανθρώπους όπως και είναι. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσω τον ε, Charles για την ε, πολύ καλή γνωμοδότησή του, η οποία καθορίζει ποια είναι τα βασικά ε, εμπόδια, τα οποία βεβαίω τα έχουμε συζητήσει και εμεί για, πολλές φορές για το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. όπω είπε και ο κύριο Βένσον, όντω αυτή η κατάσταση την μελετούμε, την συζητούμε κάθε εβδομάδα. Φτάνουν παιδιά που δεν έχουν χαρτιά, που δεν ξέρουμε από πού είναι, που δεν ξέρουμε τι ηλικία έχουν, βρίσκονται ξαφνικά στο δρόμο ή μπλέκονται σε γραφειοκρατικά γρανάζια που του παίρνει χρόνια να ξεφύγουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ανεξάρτητα από το από ποια χώρα κατάγεται το παιδί αυτό, ένα παιδί είναι ένα παιδί. Και γι' αυτό θα πρέπει να του δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ τους ασυνόδευτους ανηλίκους και, το, και τη μαφία. Τη μαφία που εμπορεύεται παιδιά και τα εκμεταλλεύεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει την προστασία που χρειάζονται τα παιδιά αυτά στο επίπεδο που του χρειάζονται. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει και ένα σωστό σύστημα υιοθεσιών στο κάθε κράτο μέλο, έτσι ώστε να αποφύγουμε παράνομε πρακτικέ ή εκμετάλλευση των παιδιών. Όπω είπε και ο Τσάλ, ε, πρέπει όντω να έχουμε συνεκτικά συστήματα, έτσι ώστε τα ε, συμφέροντα του παιδιού να διασφαλίζονται. Πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να, κάνουν, να πάρουν σωστέ αποβάσει και να αναλάβουν δράση για να δώσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση σε ε, τέτοια συστήματα για να αντιμετωπιστεί το ανθρώπινο εμπόριο. Και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Θα πρέπει να δοθεί στου ανηλίκου που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία. Πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία και διάλογο με τι χώρε προέλευση και τι χώρε διαμετακόμιση. Πρέπει να να ανοίξουμε τους διάβολους επικοινωνίας με τα, επικοινων... με τα Υπουργεία, ε, μεταξύ Υπουργείων και Βρυξελών και σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική των, ε, της επιστροφής ε, και της επανένταξης των ανεσυνόδευτων ανηλίκων, αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο όταν η οικογενειακή κατάσταση αυτού του ανηλίκου το επιτρέπει και όταν αυτό συστήνεται να γίνει. Όταν δηλαδή το παιδί αυτό θα γυρίσει σε, μια, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. θα πρέπει βεβαίως να τους ε, δίνεται και η δυνατότητα να λάβουν την ε, ηθαγένεια ε, πριν φτάσουν στην ηλικία της ενηλικίωσης. Το σχέδιο δράση της Κομισιόν για τους ασυνόδευτους ανηλίκους είναι πολύ σημαντικό φυσικά. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο αυτό δεν καλύπτει τις βασικές παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται αυτά τα ε, ανήλικα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ε, επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, αν επιθυμεί να παρέμβει. Ο κύριος Γιάννη Σαβέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους και άκουσα ενδιαφέρουσα έκθεση της κυρίας Κρίς ε, Έχει ερευνήσει εξωτικά το θέμα. Για ποιο λόγο φεύγουν τα παιδιά, μπορεί να προσπαθούν να αποφύγουν τη δίωξη, τα ανήλικα παιδιά, να επιδιώκουν καλύτερη ζωή. Πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι παιδιά και μετά το καθεστώς που τα διέπει. Αυτό είπαν πολλοί από εσά. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να επεξεργαστεί σχέδιο δράση. Έτσι η προσέγγιση θα είναι οριζοντίου φύσεως θα είδατε ότι στο σχέδιο δράσεως καλύπτονται διάφορες νομικές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί, είναι καθοδόν προς ολοκλήρωση, καλύπτονται και προγράμματα συνεργασία με διάφορους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Αυτή η δράση απαιτείται για τη μετώπιση του φαινομένου. Πολυεπίπεδη προσέγγιση από πολλούς συμμετέχοντες, από πολλούς φορείς όπως η ΜΚΟ. Έκαναν πολύτιμη έρευνα στον τομέα η ΜΚΟ. Το Σεπτέμβριο εγκρίναμε μια διάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσεως. Στην αναθεώρηση αυτή γίνεται απολογισμός των αποτελεσμάτων, δίνονται κάποιες ιδέες για το μέλλον. Αναφέρουμε την πρόοδο που επετεύχθη στο νομικό πλαίσιο το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που τελεί υπό διαπραγμάτευση, σχεδόν τελειώνουν οι διαπραγματεύσεις και οδηγία περί επαναπατρισμού, περί επιστροφής θα σας ενημερώσουμε περί εφαρμογή στο τέλος του έτους. Η οδηγία περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις για τους ε, ασυνοδεύτους ε, ανηλίκους. Η τελευταία οδηγία που υφετήθηκε ήταν η καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων και η προστασία του παιδιού είναι βασική αρχή. Διάφορε νομικέ πρωτοβουλίε ανελήφθησαν τα τελευταία χρόνια. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή αυτών. Θέλουμε να δούμε πώ θα εφαρμόσουν τα μέτρα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να δούμε αυτό πρώτα, πριν δούμε τι θα γίνει μετά. Αυτά απαντώντας τα όσα αναφέρει η τροπολογία 4. Να αναφερθώ σε πρακτικά παραδείγματα συνεργασίας. Εμπλέκομαι προσωπικά σε αυτές τις προσπάθειες. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τεχνικά ζητήματα. Ανείχνευση οικογενειών, αξιολόγηση ηλικία. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ ετούντος άσυλο και άλλου παιδιού και χαίρομαι που όλοι το βλέπουν έτσι. Η, Άσο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη Χορήγηση Ασύλου κινείται ενεργά και βοηθά τι χώρε να συνεννοηθούν επί προσανατολισμών για τα θέματα. Αλλά δεν περιορίζεται στα μέτρα στου ετούντε άσυλο. Έτσι βλέπουμε πώ το σχέδιο δράσεω συνέβαλε στην προσπάθεια που καταβάλλεται. Ενθαρρύνει πολυσχηδή προβληματισμού και πολύπλευρη συμμετοχή. Το σχέδιο δράση λοιπόν είναι καλό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν τμήμα τη μεταναστεύσεω προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα αλλάξουν τα πράγματα μετά το 2014. Καλωσορίζουμε τι προτάσει και τι πληροφορίε σα. Μετά το 2014 πιστεύουμε ότι πρέπει να εξακολουθήσουμε τι προσπάθειε. Σχέσει με τρίτε χώρε. Σημαντικότατο αυτό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα στον πολιτικό διάλογο που διεξάγει με τρίτες χώρες. Αναφερθήκατε σε βιώσιμες λύσεις, την επιστροφή των ανηλίκων. Αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Όταν όμως ε, θεωρηθεί καλύτερη λύση αυτή, η διαδικασία που ακολουθείται είναι περιπλοκότατη πρέπει να είναι θέμα ανείχνευση οικογένεια του ανηλίκου. Πρέπει να έρθει ανήλικο σε επαφή με την οικογένειά του. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό σε κάποιε τέτοιε χώρε, αλλά μπορεί να συνεργαστούν οι χώρε. Τα διάφορα προγράμματα. Υπάρχουν κάποια. Και κάποιοι πόροι. Η ενδιάμεση έκθεση του Σεπτεμβρίου συνοδευτήκε και από ένα έγγραφο εργασία μακροσκελέ. Παραθέτει πολλά προγράμματα που έχουν στόχο την πρόληψη εμπορίου ανθρώπων ενθάρρυνση βιωσίμων λύσεων, επανένταξη των ατόμων στις χώρες καταγωγής, προέλευσης. Πολλά προγράμματα, δεν τα αναφέρω όλα. Να αναφέρω πιλωτικά προγράμματα. Προκηρύχθη διαγωνισμό για πιλωτικά προγράμματα κατ' περώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για δύο χρόνια θα εφαρμοστούν τα πιλωτικά προγράμματα για να ενθαρρυνθούν καινοτόμε προσεγγίσεις με συμμετοχή πολλών φορέων, κρατών μελών, ΜΚΟ, να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα πορίσματα των ερευνών. Αυτό υπόσχεται πολλά. Ο πρώτος διαγωνισμός μόλις έληξε και αξιολογούμε τα προγράμματα. Αναφέρατε ένα θέμα για τους ανηλίκους που ξεφεύγουν, που το σκάνε από την μέρημνα. Δεν μπορούν να κρατηθούν, να, να τελέσουν υποκράτηση οι ανήλικοι, να συλληφθούν. Καμιά φορά πέφτουν στα δίχτυα διαφόρων παρανόμων δικτύων και εξαφανίζονται. Και εκεί υπάρχουν δυνατότητε συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό στρατηγική κατά του παρανόμου εμπορίου υπήρχε και συγκεκριμένη δράση προσανατολισμού στη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών προστασία παιδιών. Διότι αυτά τα παιδιά ωφελούνται από την προστασία των παιδιών. Δεν υπάρχουν μεθοριακοί έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα καλό θα ήταν να συνεργαστούν οι αρμόδιοι φορεί προστασία των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συγκεκριμένε δράσει προβλέπονται γι' αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρενς. Για να ολοκληρώσετε παρακαλώ κύριε Γκέρενς. Ναι. Νομίζω ότι στην Επιτροπή μας ε, ομόφωνα αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε πάντο δυνατόν για το θέμα αυτό. Και όταν λέω πάντο δυνατόν, αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μίλησε για το σχέδιο δράση. Αλλά σημαίνει να πάμε και πιο πέρα. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα αριθμιστικό πλαίσιο που στην πράξη θα μεταφράζει τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως συμβαλόμενα μέρη στις συμβάσει που σα προανέφερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί πρόκειται για παιδιά. Δηλαδή για ευάλωτα, άκρος ευάλωτα ε, μέλη της κοινωνίας μας, τα οποία είναι εκτεθειμένα στα πλέον αποτρόπια εγκλήματα ε, που μπορεί κανείς να, ε, να δει στην κοινωνία μας. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να σκεφτούμε το ενδεχόμενο κατάρτιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου. Ω κοινοβούλιο δίνουμε και την πολιτική όθηση, είμαστε όμως και νομοθετική αρχή, άρα πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Και να δώσουμε την πολιτική όθηση, κυρία ε, Δισπέκ με τη δική της έκθεση, είναι αρμόδια γι' αυτό, αλλά και εμείς με την γνωμοδότησή μας. Αλλά με την κυρία Κρίσπεκ, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο τι πρέπει να κάνει και η Κομισιόν, που νομίζω ότι πρέπει να είναι η ανάληψη μια πρωτοβουλίας για να ολοκληρώσει αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο. Νομίζω ότι δερμηνεύουμε αυτά τα λόγια της απόψεων συναδέλφων. Δεν ε, υποστηρίζω ότι ικανοποιεί πάντως με αυτό, Τέλο πάντων. Πρόεδρος, η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης είναι 21η Μαρτίου, 12 η ώρα. Και ψηφίζουμε 23 ε, Απριλίου, συγγνώμη. Nous allons maintenant aborder le point 8. Περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της ημερησιάς διάταξης. Ε, de notre projet d'avis. για ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, για τη σύσταση προς το Συμβούλιο για την 68η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Κρίστοφ Λίσεκ είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Θα σας δώσω το λόγο κύριε Λίσεκ για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Thank you very much, Madam Chairman. I would Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω καταρχά ότι είμαι πολύ συγκινημένο γιατί είναι η πρώτη μου γνωμοδότηση. Είναι η ιστορική λοιπόν στιγμή για μένα. Ε, για να μην ασπαταλήσω το χρόνο, βλέπετε το κείμενο της ε, γνωμοδότησης. Η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2013 και θα επικεντρωθεί κυρίως στην βιώσιμη ανάπτυξη, στους σχετικούς στόχους και στους στόχους μετά τη χιλιετία. Θα πραγματευτεί ε, θέματα όπως κράτος δικαίου, δημοκρατία, ε, ειρήνη και ασφάλεια στις ε, σε επικίνδυνες περιοχές, ανθρωπιστική βοήθεια, ασφάλεια εργαζομένων, ευθύνη προστασίας Επίσης, για την κατά μου την άποψη, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε τέσσερις τομείς. Πρώτον, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι σχετικοί στόχοι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ο σύνδεσμος μεταξύ της πρόσβασης στην ενέργεια και στο νερό, την βιώσιμη χρήση της γης, την προστασία των θαλασσών, τη βιοπικιλότητα και των φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση των της κλιματικής αλλαγής ε, είναι, ε, και, της, ε, και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικό ως δυνατότητα. Η πρόσβαση στο νερό επίσης είναι πολύ σημαντική, οι βιώσιμες υπηρεσίες ενέργειας, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις αντιμετώπισης της πείνας, η πτυτικότητα των τιμών, η ενίσχυση των, των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες περιοχές είναι επίση εξίσου σημαντικά θέματα. Δεύτερον, μετά το 2015 και το σχετικό πλαίσιο ανάπτυξη. Συμφωνώ με τον κύριο Κατσμάρα και την σχετική, ε, το σχετικό σχέδιο ε, έκθεσης ε, για το μετά το 2015. Νομίζω ότι όταν συζητούμε για την ανάπτυξη θα πρέπει όντως να επικεντρωθούμε μετά το 2015 και να πούμε ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια καθώς επίσης και την ανισότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και η σχετική προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως τη δημοκρατία ε, θα πρέπει να υιοθετηθεί. Ε, επίσης υπάρχει μεγάλη, ε, δίνεται μεγάλη σημασία στην αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη συνεκτικότητα της πολιτικής και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής βοήθειας. Επίσης, η χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει για μετά το 2015 να δώσει ένα 0,7% του ΕΠ, του καθάριστου εθνικού προϊόντος της. Αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν και αποτελεσματικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως ας πούμε οι ε, συμπράξει ε, ε, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κάποιε δανειακέ συμβάσει και τέτοιες, ε, πρόσβαση σε τέτοιου μηχανισμού από τι αναπτυσσόμενε χώρε. Επίση, ε, ειρήνη και ασφάλεια. Στην γνωμοδότησή μου τονίζω το ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ τη ανάπτυξη και τη επανένταξη, ε, να, ενισχυθεί ο συντονισμό μεταξύ ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και όσων ασχολούνται με την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόλτες Ντάστρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ουσιαστικά ε, θα πω αυτά τα οποία θα έλεγε ο συνάδελφος ε, Σαλόμεν Ενέργεια Γκερέρο που δεν μπορεί να είναι εδώ. Θέλω να σας ε, υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικές είναι οι σύνοδοι αυτοί για την αναπτυξιακή βοήθεια και ιδίως για του αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πια δεν μπορούμε ε, να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα καθώ και στο τομέα της εκρίζωσης τη στόχιας αν δεν έχουμε στο μυαλό μα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει συνένεση, πιστεύω, ευρύτατη συνένεση στη διεθνή κοινότητα από αυτού, Όμω αυτή η γενική συμφωνία θα πρέπει να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα. και δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε τους στόχους, ε, ε, ιδίως τους αναπτυχικούς στόχους της Ήλιτες 2015 θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους στόχους αυτούς ε, τις επόμενα, τα επόμενα χρόνια στην Επιτροπή μας. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το σενάριο 2015. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση, τα πεπραγμένα μέχρι τώρα, να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε και αν έχουμε αποτύχει πού και γιατί αποτύχαμε. Επίσης πιστεύω ότι αυτή όλη η συζήτηση και προβληματισμός για τους στόχους χιλίτες μετά το 2015 ε, μια διαδικασία που ξεκινάει θα πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο συμμετοχική. Θα πρέπει να συμμετέχουν όχι μόνο τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και όσο δυνατόν περισσότερε οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών και από το και από τον Νότο. Γιατί αυτό θα βελτιώσει και την ε, έννοια της, ε, και την ιδιοποίηση, την οικειοποίηση αυτή τη όλη διαδικασία. Θα πρέπει επίσης να έχουμε και ένα θεματολόγιο χρηματοδότησης ρεαλιστικό ε, με στόχους, γιατί αλλιώς η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της και κατά ποσά πιθανότητα ε, και οι προσδοκίες των πολιτών που βάζουν πολύ ε, ψηλά προτεραιότητές στην καταπολέμηση της στόχιας θα απογοητευτούν. Έχουμε μια ευθύνη λοιπόν, μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει ηγετική ε, στάση σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρενς. Έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος είπε ότι είναι η πρώτη έκθεση του που συντάσσει εντός Επιτροπής μας. Θα ήθελα να τον συγχαρώ έξοχη δουλειά. Αλλά τι θα γινόταν αν ήταν απλή γνωμονότηση με αυτή, τη, θα, με αυτή την αρχή ε, που έκανε θα, ήμασταν, θα επικρατούσε εφορία. Να πω δύο πράγματα πρώτα απ' όλα. Στην επόμενη συνέλευση, θα πρέπει η επόμενη συνέλευση του ΙΕ να είναι χρήσιμη. Και η Επιτροπή που μπόρεσε να τοποθετηθεί εκεί έδειξε ότι έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Ελπίζω ότι η Πίμπαλξ να μπορέσει να αφήσει το ίχνος του στην επόμενη σύνοδο ε, είμαστε οι πρώτοι ε, χρηματοδότες δανειστέ. Εμείς πρέπει να είμαστε σημείο αναφορά για όλους και για τα Ηνωμένα Έθνη σαν θεσμό, διότι χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που είναι πρώτο δωρητή, ο ΙΕ θα ήταν καταδικασμένος σε ανυπαρξία. Ή θα είχαν μειωθεί κατά πολύ οι φιλοδοξίες του ΟΗΕ, κυρίως στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε στην ευθύνη όλων, να την επικαλεστούμε. Και θα είναι και η πρώτη δοκιμή για την διαφοροποίηση, για την έννοια αυτή. Αν θέλουμε να πετύχουμε τις, τους αντισιακούς στόχους της χιλιετίας, αν θέλουμε μετά το 2015 ε, να πετύχουμε αποτελέσματα σε σχέση με τους αντισιακούς στόχους της χιλιετίας, ε, θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε κατάλληλα. Πρέπει να κινηθούμε σοβαρά, δεν θέλουμε ιστορίες και διασκέδαση. Εκείνοι που παράγουν τα διάφορα μέσα θα πρέπει να τα εφαρμόζουν σωστά για να καταπολεμηθεί η ένδια. Κατά είμαι, είμαι κατά παθού τοποθέτησης τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στη Νέα Υόρκη. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία και θα πρέπει να βασιστούμε στην, στα, στα πορίσμα της του συναδέλφου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω να μπορεί να, να εκείνοι που θα παραστούν στις συζητήσεις ε, στη Νέα Υόρκη θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν κάπως τα τεκτενόμενα στις συζητήσεις στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για ένα λεπτάκι μόνο. Η έκθεση που μας παρουσιάζει ο συνάδελφός είναι καλή, ευφύης, σύντομη και συγκεκριμένη, ακριβής έκθεση. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν κατάλογο πιθανών συμβιβασμών. που ότι θα πρέπει ο εισηγητής της έκθεσης να τις λάβει υπόψη του τις προτάσεις αυτές. Αυτά που λέει ο κύριος Γκέρνς, τώρα δεν ξέρω αν είναι επίτροπος. γιατί δεν μιλά ε, στην Ολομέλεια των Εθνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, νομική προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν είναι ο επίτροπος δηλαδή αυτός που θα μιλήσει ή ή κάποιος ε, υψηλότερος αξιωματούχος. Συμφωνώ πάντως με αυτά που είπε ο κύριο Γκένος ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά νομίζω ότι η έκθεση που μας παρουσίασε ο συνάδελφος Λίσεκ είναι φιλόδοξη γιατί είναι πολύ ακριβή, συγκεκριμένη. Ίσως είμαι ο βετεράνος εδώ στην ομάδα. Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν κύριε Λίσεκ και να σας πω ότι για δεκαετίες χρησιμοποιούσαμε την έκφραση χάνω την παρθενιά μου. Αλλά μάλλον δεν πρόκειται γι' αυτό. Μιλάμε πιο πολύ για το ότι ανεβαίνουμε επίπεδο. Περνάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό κάνατε κι εσείς. Αφήσατε την ε, παρθενία σας εντός αγωγικών αφού πλέον γίνεστε συντάκτης έκθεσης. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μπάρμπαρα Λουέκ, και ο κύριος Πέντρο Ενρίκες την εκπροσωπούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, και συνάδελφος πρέπει να είναι εδώ. Συνεργαζόμαστε στενά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους συναδέλφους τους αρμόδιους. Θέλουμε να περιορίσουμε τα σχόλιά μας όσον αφορά το αναπτυξιακό τμήμα της συζητήσεως. Θα έλεγα ότι η 67η Σύνοδος του ΟΗΕ, της συνελεύσεως, ε, τα πορίσματα της Γενικής Συνελεύσεως αποτελούν προτεραιότητες. Όμως, η 68η Σύνοδος ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη. Έγιναν συζητήσεις για το τι θα γίνει μετά το 2015 Διάφορα αναθεωρήσεις πρέπει να γίνουν, Δραστηριότητε θα ακολουθήσουν. Ρίο συν 20 διάσκεψη, τη συνέχεια θα δοθεί. Το υψηλού επίπεδου πολιτικό φόρουμ που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στο ΟΝΚ 68, στην 68η Σύνοδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και έχουμε και ομάδε εργασία που ασχολούνται με του στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη χρηματοδότηση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αθέτησε πρόσφατα μία ανακοίνωση. Αξιοπρεπή ζωή για όλου είναι ο τίτλο τη. Προτείνεται κοινή προσέγγιση ευρωπαϊκή για τα θέματα. Κάτι μπορεί να συμβάλλει να συγκεράσει τι διαδικασίε του ΟΗΕ για μία ανάπτυξη μετά το 2015. Μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο. Βλέπετε τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα αύριο, που προβλέπονται. Με τις συζητήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα σχετικά με το τι προσεγγίσεις θα ακολουθούν μετά το 2015. Βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται μια πιο γενικόλογη παράγραφος. Θα αναφέρεται στην ανάγκη αποτελεσματική συμπερίληψη των τριών διαστάσεων της βιώσιμης αναπτύξεως. Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τέτοια. Θέλουμε αποτελεσματικότερη εφαρμογή στον ΟΗΕ. Χρηματοδότηση αναπτυξιακή. Χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση. Βάσει των συζητήσεων. Χρηματοδότηση και μέσα εφαρμογή των πορισμάτων και του ριου και των συζητήσεων για το κλίμα και άλλων συζητήσεων. Χρειάζεται σφαιρική, ολιστική προσέγγιση στον τη χρηματοδότηση χρηματοδότηση δημόσια, ιδιωτική, κρατική, διεθνής, εσωτερική, ιδιωτική χρηματοδότηση, προτεραιότητες, έλεγχος, Η διεθνής μετανάστευση και ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γίνονται συζητήσεις σε ψηλό επίπεδο σχετικά με αυτό. Τον Οκτώβριο του 2013 θα γίνει η συζήτηση υψηλού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει σχετική ανάπτυξη. Τίτλο Βελτιστοποίηση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων της μετανάστευσης. Στόχος της ανακοίνωσης να συμβάλλει στην καθιέρωση της θέσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις συζητήσεις του ΙΕ σε υψηλό Να διερευνήσουμε επίσης τα επόμενα βήματα για τη συζήτηση του θέματος των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων της μετανάστευσης. Ένας επιτυχής διάλογος σε υψηλό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει τη γενική συζήτηση για τη μετανάστευση και για την ανάπτυξη. Αυτά είναι τα σχόλια. Ε, merci Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λίσεκ για να καταλήξει. Thank you very much, Madam ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω Επιτροπή ανάπτυξη, βεβαίω εμεί θα συζητήσουμε για την ε, γνωμοδότηση, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί είμαι και πλήρη μέλο στην ε, ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λοιπόν, να δεχτούν και οι συνάδελφοι από την ΑΦΕΤ την γνωμοδότησή μας. Θυμάμαι από το παρελθόν, όταν συμμετείχα σε, στην αντιπροσωπεία της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παρόλο που δεν είμαστε πλήρη μέλη, θυμάμαι ότι ως αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε πολλές συναντήσεις με σημαντικούς ανθρώπους, με τον πρόεδρο ας πούμε, της ε, Γενικής Συνέλευσης ε, στη Νέα Υόρκη και με άλλους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από όποιον πάει, εκπροσωπώντας ε, το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τους συναδέλφους να πάρουν την γνωμοδότησή τους και την έκθεση της ΑΦΕΤ και να την προωθήσουν στους, σε όσους συνομιλήσουν είναι νομίζω σημαντικό να το κάνουμε αυτό στη Νέα Υόρκη ως ε, κοινοβούλιο, ως ε, αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και βεβαίως ευχαριστώ και όλους τους ε, συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για τα καλά τους λόγια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για αυτή τη γνωμοδότηση λήγει στις 26 Μαρτίου 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε 23 Απριλίου. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 9 της Μέσας Διάταξης που έχουμε να ακούσουμε την ε, παρουσίαση για την, επιτροπ... την ε, αποστολή φυλακής παρατήρησης της Χέρα Λεόνε. Ο συνάδελφος ε, Τσαρτ Χάουιτ ήταν ο επικεφαλής της αποστολής παρατήρησης. Θα σας δώσω το λόγο κύριε Χάουιτ για να ακούσουμε τον απολογισμό της αποστολής σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντα πόσο χαίρομαι που επέστρεψα στην Επιτροπή Ανάπτυξη εδώ. Πέρασα εννέα χρόνια ευχάριστα σε αυτή την Επιτροπή σαν μέλο και τώρα εστιάζομαι στην, σε έργο τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικοδόμηση δημοκρατία και είναι μεγάλη χαρά που παρουσιάζομαι εδώ. Συνεργάζομαι με πολλού φίλου αυτή τη Επιτροπή και ελπίζω ότι κάποια μέρα ίσω να επανέλθω, αν με δέχεστε. Επίση, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά την εμπειρία που είχα που ήμουν επικεφαλής των παρατηρητών των εκλογών. Ξανά είχα το προνόμιο αυτό να είμαι παρατηρητής εκλογών για δέκατη φορά εκπρόσωπος αυτού του κοινοβουλίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εδιορίστηκα επικεφαλής παρατηρητής και είναι απίστευτο προνόμιο για ένα Ευρωβουλευτή να αναλάβει αυτό το ρόλο και είμαι βαθύτατα υπερήφανος για την ομάδα την εκατονταμελή των ε, παρατηρητών που εκπροσωπούσαν 26 χώρες και είμαι περήφανος και για το έργο της αποστολής μας και θα ήθελα να πω ότι η βασική ομάδα και οι παρατηρητές των εκλογών ήταν με... Ήταν πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και θέλω να επενέσω επίσης και τη συνάδελφο Μαρία Γκάμπριελ και τους άλλους ευρωβουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή. Τους ευχαριστώ βαθύτατα, ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν και πάνω απ' όλα την ίδια τη χώρα που μας προσεκάλεσε να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο. Η Σιέρα Λεόνα είναι η χώρα που είναι στο κατώτατο σημείο του πίνακα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και όταν σας το λέω αυτό ότι από μια ομάδα 30 μακροχρόνιων παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, 11 τουλάχιστον έπρεπε να απομακρυνθούν διότι έπαθαν είτε τυφοειδή πυρετό ή ελονοσία και πρέπει να δείτε πόσο μεγάλη είναι η φτώχεια της χώρας και ήρθε και σε εμά, στο σπίτι μα, στου Ευρωπαίου, με έναν τρόπο που αποτελεί πραγματικότητα καθημερινή για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή... της ε, Λεόνε. Ήδη συνέταξα μια έκθεση και κλεισμένων των θυρών, την υπέβαλα στην ομάδα συντονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη τη δημοκρατία και για τι εκλογέ. Δεν θα επαναλάβω τώρα εκτενώ τι λεπτομέρειε, αλλά στην τελική έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στην αίθουσα ε, και online, αναφέρονται αυτά. Θα προσπαθήσω στα σχόλιά μου σήμερα το απόγευμα να εστιαστώ επί κάποιων γενικών συμπερασμάτων που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του έργου που επιτελεί σε συνεργασία με αυτή τη χώρα και τώρα και στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, ε, σαφώς ήταν εκλογές που έλαβαν χώρα μετά την σύραξη. Είναι οι τρίτες εκλογές μετά τον αιματηρό και βίο ε, ε, φίλιο πόλεμο της Σιέρα Λεόνη και όλοι είπαν ότι η πρόκληση αυτή των εκλογών θα ήταν κατά πόσο η χώρα θα μπορούσε να δείξει ότι μπορεί να μετακινηθεί από μια μεταπολεμική ε, εποχή σε μια αναπτυξιακή φάση. Αυτό δεν εναπόκειται σε εμά που είμαστε παρατηρητέ των εκλογών να το συμπεράνουμε. Αλλά είπαμε στην αρχική μα δήλωση ότι οι εκλογέ αυτέ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια δημοκρατική εξυγίανση και αυτό θα μπορούσε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη χώρα και στη διεθνή κοινότητα αυτή η λέξη ότι θα μπορούσε να οδηγήσει, δημιουργεί το κλίμα είναι σημαντική, διότι σημαίνει ότι είναι δυνατόν, εφικτόν, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Ε, δεύτερον, σαν μέλη αυτή τη επιτροπή, ε, τα μέλη αυτή τη επιτροπή θα το καταλαβαίνουν, ενώ αυτοί που είναι απ' έξω δεν το καταλαβαίνουν, βασικό θα ήταν να δούμε κατά πόσο η σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων και των υποστηρικτών του θα οδηγούσε στη βία Δυστυχώς υπήρξαν κάποια επεισόδια βία, ε, μαχαιρώματα, απαγωγές, σεξουαλική βία, λιθοβολισμοί, εμπρισμοί ε, και περιπτώσεις διατάραξης της τάξης θα μπορούσε να πει κανείς. Ε, όμως αυτά τα επεισόδια ήταν σποραδικής φύσεως, δεν έγιναν ανεξέλεγκτα και η μεγαλύτερη δοκιμή όλων, κανένας δεν πέθανε. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι οι εκλογές ε, ήταν γενικά ειρηνικές και εκστρατείε καταπολέμησης τη βία συνέβαλαν τα μάλα από το αποτέλεσμα και εμείς προτείνουμε τη συνέχιση των μέτρων οικοδόμηση εμπιστοσύνη αμέσω μετά. Αλλά οι ηγέτες των κομμάτων έδωσαν υποσχέσεις και τι ετήρησαν και θα πρέπει να τύχουν συγχαρητηρίων γι' αυτό και αυτοί που έχασαν τις εκλογές και αυτοί που νίκησαν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε με τη σωστή ταπεινότητα όπως μας είπαν πολλοί άνθρωποι της Ιερα Λεώνα, ότι η παρουσία μας σαν αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοήθησε να τους δώσει εμπιστοσύνη όσον αφορά την εκλογική διαδικασία και έτσι μπόρεσε εν γέννη να είναι ειρηνική αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει καλύτερη μαρτυρία όσον αφορά το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, υπήρχαν κάποια σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ε, διεξαγωγή των εκλογών στην έκθεση. Είπαμε ότι δεν ήταν ισότιμες συνθήκες και αυτά είναι κενά τα οποία θα πρέπει και μπορεί να τα καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, δεν μπορούσε να σημειωθεί καμία πρόοδο όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών. Ένα από τα κενά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ενίσχυση ε, την παιδεία των εκλογέων και όσον αφορά την αγωγή του πολίτου λόγω τη ε, αγραμματοσύνη στη χώρα και θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει στο δικαστικό τομέα, τους, ώστε οι εφέσει ε, και οι καταγγελίε να γίνονται έγκαιρα και να επιλύονται, κάτι που δεν έγινε τώρα, για να μην επηρεάζονται εκλογέ. Και θα πρέπει να θεσπιστούν και διάφορε νομοθεσίε για τη διαφάνεια τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, συνομίλησα με τους πρεσβευτές των κρατών μελών ε, στο Freetown και με τους έξοχους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τη αντιπροσωπεία εκεί, συζήτησα εκτενώς και καταλήξαμε σε κάποιες συστάσεις αναποστολή συγκεκριμένε και πρακτικές που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ε, ε, όσον αφορά την υποστήριξη που χορηγείται ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το 11ο, το 11ο Αναπτυξιακό Ταμείο Λοιπόν, ζητούμε από τον Επίτροπο της, ε, τον και αυτή την Επιτροπή να εστερνιστούν αυτές τις συστάσεις ε, ούτως ώστε τελικά να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι προσπάθειές μας. Όλοι να γνωρίζουν ότι με τέτοια συνέχεια μετά τις αποστολές παρατηρήσεων εκλογών είναι κάτι καταρχήν σωστόν. Και στην περίπτωση της Ιερα Λεώνα ελπίζω να αποτελέσει υπόδειγμα σχετικά με το πώς αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη. Τέταρτον, έγινε σημαντικό βήμα προόδου προ ανάπτυξη όσον αφορά αυτές τι εκλογές. Οι πρώτερες εκλογές ουσιαστικά διεξήχθησαν από τον ΟΗΕ και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο χώρο του ε, Βρετανικού Συμβουλίου της ε, Freetown. Αυτή τη φορά οι εκλογές ε, καθοδηγήθηκαν από τι αρχές Λεώνα και πρωταρχικό λόγο είχε η Επιτροπή Εκλογών Ιερα Λεώνα και η ίδια Διευθύνουσα Επιτροπή τη Κυβερνήσεω διεξήγαγε τι εκλογέ. Ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, τώρα είναι Υπουργό Εξωτερικών, που ηγήθηκε τι προσπάθειε. Βασική υποστήριξη έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δώσαμε χρήματα για την οικοδόμηση δημοκρατία, ένα τρίτο του συνολικού κόστου των εκλογών χρηματοδοτήθηκε από αυτό και μέσω του έργου του ΟΗΕ και των τεχνικών συμβούλων τη Νιγηρία χορηγήθηκε βοήθεια. Όμω ήρθαν ε, τα διάφορα παραβάν όσον αφορά τι εκλογέ από την Κάνα και τα διάφορα ψηφοδέλτια τυπώθηκαν στην Νότια Αφρική. Και όσον αφορά το ρόλο μα, σαν παρατηρητέ συνεργαστήκαμε με του ντόπιου ε, παρατηρητέ και με διάφορε ομάδε από την ECOWAS, την Κοινοπολιτεία και την Αφρικανική Ένωση. Και πιστεύω ότι μάθαμε σημαντικά μαθήματα σχετικά με το πώ μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά αποτελεσματικότερα στο μέλλον. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η συνεδρίαση θα καλωσορίσει τι καλέ αναπτυξιακέ αρχέ που ε, ε διέπνευσαν την προσπάθεια μα, που θα πρέπει βέβαια να είναι σημαντικό τμήμα των διαφόρων αποστολών για τις εκλογές στις διάφορες αναπτυσσόμενε χώρε. Και τέλο, εν μέρη σε αυτό το πλαίσιο, έχω ένα βασικό μήνυμα το οποίο μπορώ να συναγάγω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτή την Επιτροπή, καθώ και για τη διεθνή κοινότητα γενικότερα. Η Σιέρα Λεόνε είναι μια χώρα όπου έγινε η πρώτη ποτέ ε, ειρηνική μετάβαση, ε, μεταβίβαση εξουσίας οπουδήποτε στην υποσαχάρη Αφρική. Είναι σημαντικό εντός της χώρας αλλά και εκτός αυτής οι συνθήκες για παρόμοια μεταφορά της εξουσίας και σε τωρινές και σε μελλοντικέ εκλογές να παραμείνουν, να ισχύσουν ε, και υπάρχουν και κάποια μηνύματα προειδοποιητικά. Η υποστήριξη για τα δύο βασικά κόμματα παρέμεινε εδρασμένη επιθνωτικών διαρέσεων και αντικατόπτριζε και περιφερειακές υποδιαρέσεις στη χώρα και η πόλωση φαίνεται ότι αυξανόταν σε αυτές τις εκλογές. Ε, παρατηρήσαμε πολύ χαμηλά επίπεδα εκστρατιών διότι πολλά καταχωρημένα πολιτικά πέρα από τα άλλα πολιτικά κόμματα, πέρα από τα βασικά κόμματα, άρα χαμηλό ο ανταγωνισμό στι εκλογέ. Παρεμποδίστηκε. Δεν δόθηκε ιδιαίτερο τότε σε άλλα κόμματα και υπήρχε σημαντική ανισορροπία στα μέσα ενημέρωσης και κακή χρήση επίσης των κρατικών πόρων. Και αυτά συνέβαλαν στο να υπάρχει ανισορροπία και αδικία στον αφορά την προηγική εκστρατεία. Αν τα βάλουμε όλα αυτά σαν παράγοντε μαζί, συμπεραίνουμε. Και θέλω να πω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την ενασχόλησή τη, να συμμετέχει περισσότερο στι διεργασίε στη χώρα. Και είναι πολύ πιο σημαντικό αν υποβαθμίσει ο ΙΕ τι δικέ του δραστηριότητε εκεί το επόμενο 12 μήνο. Σε μια περίοδο περιορισμένων πόρων παραδέχομαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε να κάνουμε η δημοκρατία και για την ανάπτυξη παντού. Όμως ε, η Σιέρα Λεόνε είναι μια χώρα όπου η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα έχει επενδύσει πάρα πολλά στην ε, μεταπολεμική ε, εποχή. Μια χώρα που είναι ανοιχτή και δέχεται διεθνή υποστήριξη και βοήθεια. Μια χώρα που πιστεύω είναι μια επιτυχία ε, για την διεθνή κοινότητα και πάνω απ' όλα για την ίδια τη Σιέρα για το λαό τη Σιέρα Λεώνα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το αναποφευτό όσον αφορά την παραμονή της ειρήνης και της δημοκρατίας και όταν ε, συζητείται εκτενώς το πώς πραγματικά μπορούμε να μειώσουμε ε, τους πόρου πόρους μετά την στατιωτική παρέμβαση σε χώρες αλλαχού στον κόσμο, η Σιέρα Λεόνα είναι μια χώρα όπου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο αυτό το θέμα, πώς θα μειώσουμε τους αναπτυξιακούς μας πόρους, έχοντα ε, έχοντας υπόψη τον ίδιο στόχο, ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να παραμείνει η ειρήνη και η δημοκρατία στη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η Επιτροπή που συζητά αυτές τις προκλήσεις, θα τις συζητήσει μάλλον, και είμαι ευγνώμων που έχω τη δυνατότητα σήμερα να συμβάλλω στη συζήτηση σας. Σας ευχαριστώ. Μαντάμ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκαμπριέλ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να επικροτήσω το έργο του κεφαλής της αντιπροσωπείας ε, των παρατηρητών και τη δουλειά που κάναν όλη, όλη η ομάδα των παρατηρητών στη Σιεραλεόνε. Θέλω να εκφράσω επίσης τι ευχαριστίες μου και στην Επιτροπή Εκλογική Παρατή και στο ΣΥΟ για το ότι μας υποδέχθηκαν πάρα πολύ καλά εκεί. Ενσωματωθήκαμε στην αποστολή παρατήρηση των εκλόγων και συμφωνούμε και απόλυτα με τα πορίσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρατηρήσαμε πολλά χαρακτηριστικά ε, στοιχεία για αυτή τις εκλογές. Πρώτα απ' όλα ήταν ειρηνικέ εκλογές, έλειπε ε, η βία. Αυτό το είπε και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο επισημάναμε ήταν τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν. Ήταν τριπλή η ψηφοφορία και έπρεπε να διδαρματίσει κεντρικό ρόλο η Εθνική Εφρευτική Επιτροπή. Κάτι που μας ξέπηξε θετικά επίσης ήταν η ενεργό συμμετοχή αφενός του συνόλου του πληθυσμού. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν του, της τάξης του 83%. Μακάρι να το είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Όνειρο είναι για μας. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα με τα μέσα που έχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να βελτιωθεί. Όλοι μας διαπιστώσαμε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μια σαφής νομοθεσία για τη χρήση κρατικών πόρων. Είδαμε ότι υπήρχε μεροληψία υπέρ κάποιων κομμάτων. Επίσης, έχουμε τομείς κλειδιά όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση, η παιδεία που πρέπει να έχουν οι ψηφοφόροι, η αγωγή, ας πούμε, πρέπει να δοθεί στους ψηφοφόρους. Ε, όλα αυτά πρέπει να, να υποστηριχθούν οικονομικά. Επίσης, συμμετοχή γυναικών, πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, αλλά για μας είναι μια θεμελιώδης αξία η συμμετοχή των γυναικών και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσα, έχει τρόπους για να συνεχίσει να προβαίνει σε θετικές ενέργειες και να παροτρύνει την κυβέρνηση να βάλει τις γυναίκες σε πόστα λήψη αποφάσεων. Θέλω επίσης να επιμείνω στην παρακολούθηση. Στη συνέχεια μπορεί να δοθεί Συμφωνώ, επαναλαμβάνω, με τα πορίσματα της Επιτροπής και της Αποστολής Παρατήρησης. Ο συνάδελφος ε, Ρικάρντο Κορτές Λάστρα είναι εδώ. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως και όλα τα μέλη της Αντιπροσωπής του Κοινοβουλίου που συμμετείχαν εργά στην Αποστολή. Να ευχαριστήσω τον επικεφάλη της Αντιπροσωπείας που μας επέτρεψε να ζήσουμε μαζί του αυτή την καταπληκτική εμπειρία και συμφωνώ μαζί του προς το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα έχει να κάνει πολλά στη χώρα αυτή με την προπόθεση η πολιτική πτυχή, ο πολιτικό διάλογο να συνοδευτεί και από συγκεκριμένα μέτρα στον οικονομικό τομέα, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντεκάιζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη χαρά τους δύο επικεφάλεις αντιπροσωπείας τελικά, τις πιο ε, και τις λιγότερο. Ε, μακροχρόνιας, δηλαδή ε, αυτής της Ένωσης και της άλλης του Κοινοβουλίου για τις εκλογές τη της Χέρα Λεόνε. Και στη Μαρία και στον Ρίτσαρτ θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Τι βλέπετε. Για, ε, τι συνέχεια συγκεκριμένη πρέπει να δοθεί δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Εδώ και χρόνια, ουσιαστικά και από την προηγούμενη θητεία, συνέχεια κρούω τον κόδωνα το κινδύνου, το συναγερμό. Ε, σημαίνω για το τι μπορεί να σημαίνει ότι εμφανιζόμαστε μεν στις εκλογές, αλλά μετά εξαφανιζόμαστε. Αυτό έχει ξαναγίνει. Το είπαμε και με τους συναδέλφους από τον Νότιο Σουδάν το μεσημέρι, με το που θα βγει από τις προβολείς ε, μια χώρα, ε, χάνεται, χάνεται. Είμαστε ίσως αρκετά παρόμοιοι με κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που με το που θα σβήσουν οι προβολείς δημοσιότητας δεν ασχολείται κανένας. Ε, πρέπει να κάνουμε πολλά λοιπόν και σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο, στον κοινοβουλευτικό διάλογο κτλ, Συγκεκριμένε δράσεις. Ένα γενικό σχόλιο ήταν αυτό τώρα. σου πω στον Ρίτσαρντ που μας μίλησε για μια πολύ εύθραυστη δημοκρατία μετά από την ε, σύγκρουση. Επειδή μιλάμε για συγκεκριμένε δράσει. εσύ τι βλέπει, Ρίτσαρντ συγκεκριμένα, τι βλέπετε εσείς οι δύο συγκεκριμένα αφού ήσασταν εκεί. Τι ιδιομορφή έχει αυτή η χώρα ε, που δεν υπάρχει κάπου αλλού. μπορούμε να πούμε ναι, θα στείλουμε βουλευτέ να έχουν συζητήσει κτλ. Αλλά εγώ αυτό που δεν ε, καταλαβαίνω πολύ καλά, γιατί δεν γνωρίζω πολύ καλά τη χώρα, είναι τι συγκεκριμένα για τι Γεραλέων θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ κύριος Κορτές Λάστρα, είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα αφήσω ή στον συνάδελφο Ρίτσαρτ Χάουιτ ή στην ε, Μαρία να απαντήσουν στο ερώτημα της Βερονίκ και ίσως να σχολιάσω εγώ μετά. Θέλω να συγχαρώ τον Ρίτσαρτ Χάουιτ. Ήταν καταπληκτική δουλειά του. Ειλικρινά είμαστε όλοι περήφανοι ε, για το έργο που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε μια πολύ δύσκολη, πολύπλοκη χώρα. Και ούτε ήταν ε, ξεκάθαρο τίποτα. Με την πρώτη ψηφοφορία δεν υπήρχε πλειοψηφία και φοβόμαστε μήπως υπάρξει ε, πρόβλημα και σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ο ρόλος των γυναικών, τη συμμετοχή των γυναικών, πράγματι όλοι μας συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών, ιδίω στη χώρα αυτή της Χεραλεόνη. Δεύτερον, εμείς ε, πήγαμε γύρω εκεί στη Freetown, στην Ήπεθρο, ε, ε, στις αγροτικές περιοχές. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έγιναν πολλές συνεντεύξεις τύπου, όμως η σημαντικότερη, Ρίτσαρτ, ε, συνέντευξη τύπου, ήταν αυτή που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έδωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια ήρθε και το έδρυμα Κάρτερ μετά και τα λοιπά τέλος πάντων, αλλά αυτό λέει πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα ε, για τη δέσμευση μετά. Υπάρχουν οργανώσεις με τις οποίες εμείς συνεργαζόμαστε συντονισμένα μπορούμε κατά. Πάντω, η ε, πιο άρθρη παρουσία ήταν στην συνέντευξη τύπου που, που έδωσε ο Ρίτσαρτ τώρα για του δύο υποψηφίου κτλ. Είδαμε την τεράστια αυτή συμμετοχή, το είπε η Μαρία. Είχαμε και ε, σε κάποια εκλογικά τμήματα κάποιε νυχτερινέ ε, Και το βράδυ η καταμέτρηση των ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα γιατί ήταν γεμάτα ε, από ψηφοφόρους μέχρι αργά. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει τις δεσμεύσεις μας να τις διατηρήσουμε, αλλά και να τις αυξήσουμε ακόμη περισσότερο. Ε, ολοκληρώνοντας να συγχάρω για μια ακόμη φορά τους δύο συναδέλφους, τον Ρίτσαρτ και την δική μας επικεφαλής αντιπροσωπής του Κοινοβουλίου. Γιατί είμαστε λίγες μέρες, πολύ λίγες, ε, αλλά Είδαμε ψοψηφίους, ε, δημοσιογράφους, ε, εκπροσώπους κοινών των πολιτών. Ε, πάρα πολλά άτομα είδαμε. Είδαμε ότι υπήρχαν προβλήματα. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που μόλις έβγαινε από σύγκρουση και πραγματικά εντό αγωγικών ομαλά κύλησαν όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκέρενς, το Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της και Κεζέρ για την ε, συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί. Όταν, ε, είμαστε, όταν ε, έχει εκλογές είμαστε παρόντες, ενώ μεταξύ των εκλογών είμαστε απόντες. Ένα κοινοβούλιο όμως εκλέγεται για να έχει κάποια δικαιώματα και καλό είναι να παρακολουθούμε αν μπορεί να τα επιβάλλει αυτά τα δικαιώματα ή να γίνουν σεβαστά, τέλος πάντων, το κοινοβούλιο. Έχουν τα κλεμμένα κοινοβούλια δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και για την παρακολούθηση, για τη συνέχεια που μπορούμε να δώσουμε, ε, θα πρέπει να ε, πούμε τα εξή. Θα πρέπει να δούμε αν έχουν έλεγχο επί των οικονομικών υποθέσεων. Έχουν μήπως ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια ή το Εθνικό Κοινοβούλιο εκεί τι ίδιε αρμοδιότητε που έχουμε εμεί, ε, παραδείγματο χάρη στο Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Γιατί αν είναι τόσα τα δικαιώματα τόσο τα δικά μα, δεν είμαστε ενώπιον μια τέλεια δημοκρατία. Εντάξει, το λέω σα αστείο βέβαια, αλλά, ε, ω ανέκδοτο, αλλά ε, τούτο λεχθέντο η εκλογική παρατήρηση μα ε, διδάσκει κάποια πράγματα. Και είναι σημαντικά αν ήταν η προεκλογική εκστρατεία σωστή, αν υπήρχε πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν τα συναγωνιζόμενα κόμματα ε, αντιμετωπίστηκαν ισότιμα, μήπως ε, ε, το κυβερνών κόμμα, η εξουσία καταπιέζει ουσιαστικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το να προβάλλεται δηλαδή συνέχεια καταπνίγονται τα άλλα κόμματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και ε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για το δημοκρατικό έλεγχο, τον έλεγχο των δικαιωμάτων. Γιατί γι' αυτό εξελέγησαν εκεί οι άνθρωποι στο Κοινοβούλιο. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω την πολύ μεγάλη αξία της δουλειάς του κύριου Χάουιτ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στις υπηρεσίες της ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ο τον Μάρκο πρόσωπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβουμε τα όσα μας είπε ο κύριος Χάουιτ. Επιβεβαιώνουμε ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συμμερίζεται απόλυτα τα όσα αναφέρθηκαν και τις εκθέσεις που συνετάχθησαν και υπευλήθησαν. Η αποστολή παρατήρηση των εκλογών εξετιμήθη τα μάλα. Όχι μόνο από τους διεθνείς φορείς, αλλά και από όλους τους εθνικούς φορείς της Ιερα Και αυτό είναι κάτι που ισχύει ιδιαίτερα στη Ιερα Λεόνε, παραπάνω από τις άλλες χώρες. Πραγματικά ήταν ένας παράγων ειρήνευσης αυξάνοντας το επίπεδο αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας ήταν ρόλο όχι μόνο παρατήρηση αυτό που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ενεργός ρόλο ε, ειρήνευσης. Εν γέννη οι εκλογές ε, καταλήγουν στα θετικά αποτελέσματα. Υπογραμμίζει όμως η έκθεση ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, τα οποία μπορούμε να συνοψίσουμε με το αν είσαι συνθήκες, αν είσαι όροι του παιχνιδιού των εκλογών. Εκεί αυτό δώσουν ο τίτλο, συμπεριλαμβάνονται διάφορα προβλήματα. Και ποια συνέχεια θα δοθεί. σα διαβεβαιώ ότι η εξωτερική υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πολιτικού διαλόγου θα δώσουν συνέχεια. Ε, επισήμως είναι στις ημερήσιες διατάξεις διαφόρων συνεδριάσεων του πολιτικού διαλόγου που διεξάγεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Σιέρα Λεόνε αυτό το θέμα και είναι και αφετηρία για τη διαμόρφωση του ενδεκάτου προγράμματος αναψυχιακής βοήθειας για την υποστήριξη της διακυβέρνησης κλπ. Κάτι που θα συζητηθεί με τους ε, εθνικούς φορείς Αυτά είχα να πω ε, όσον αφορά την πλευρά μας, την πλευρά της υπηρεσίας μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Χάουιτ, ούτω ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση, ευχαριστώνταν, το, ευχαριστώνταν, ευχαριστώνταν τον για το έργο του. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους ε, και βεβαίως όλους τους ε, ευρωβουλευτές. Πραγματικά ήταν, ήμασταν πολύ καλή ομάδα και χαίρομαι που μπορέσαμε να τα καταφέρουμε τόσο καλά. Ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε και στο μέλλον. Όταν λέτε ότι πρέπει να επιμείνουμε. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή ακριβώς είναι η Επιτροπή που μπορεί να επιμείνει και να παρακολουθήσει και να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία γιατί εμείς ως Κοινοβουλίο μέσω της Επιτροπής σας έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα όσα είπατε. Για να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε η Βερονίκ. Στην παρουσίαση μου έδωσα κάποια παραδείγματα συγκεκριμένων ελλείψεων στην όλη διαδικασία, δεν θα το επαναλάβω, αλλά οι τρόποι με, τον οποίο μπορούν, με τους οποίους μπορούν να λυθούν είναι, ας πούμε, ε, οι στεγματικές ε, αλλαγές. Ε, χαίρηκα πολύ όταν ο πρόεδρος μετά τις εκλογές ήταν σαφής που είπε ότι έχουν δεσμευθεί να το κάνουν αυτό και έχουν και δύο, άλλα δύο χρόνια για να τα καταφέρουν ε, αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία που μπορούμε να τη βοηθήσουμε και εμεί και εκεί πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Βεβαίω υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, δεν θα μπω τώρα σε παραδείγματα, αλλά υπάρχει μια πολύ καλή ε, ιστορία επιτυχία που είναι οι βιομετρικές φωτογραφίες, που ήταν πραγματικά ιδιαίτερως ασφαλείς ε, στη χρήση του. Βεβαίω, ε, δεν ε, ήρθαν όλε οι ανησυχίε για το πόσο διαφανή ήταν η όλη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι το αρχείο που δημιουργήθηκε με τι βιομηχανικέ φωτογραφίε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώ προχωράει η όλη διαδικασία προ τα Εμπρό. Γιατί βεβαίω το θέμα δεν είναι να υπάρχει μόνο διαδικασία, είναι να διατηρηθεί και σε ένα βάθο χρόνου. Και επίση υπάρχει και ένα θέμα με την εξέλιξη των κομμάτων. Βεβαίω η δημοκρατία χρειάζεται κόμματα, κανεί δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι η, τα θεμέλια της δημοκρατίας είναι πολύ πιο παρόντα στις ευρωπαϊκές χώρες, ε, στην ε, κεντρική Ευρώπη, ε, στην Ανατολική Ευρώπη ακόμα, σε σχέση με το πώς είναι η κατάσταση στις χώρες της Αφρικής. Πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε να ενισχύσουν αυτά τα δημοκρατικά θεμέλια, να δημιουργηθεί ένας ευγενής ανταγωνισμός και αυτό νομίζω ότι είναι δυνατό στη Σιέρα Λεόνε. Μπορούμε λοιπόν να τους δώσουμε κάποια κίνητρα, ίσως και χρηματικά, να ενισχύσουμε την όλη διαδικασία δημιουργίας των και εγκαθίδρυσης των κομμάτων. Τώρα πώς είναι διαφορετική αυτή η χώρα από άλλε. είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω. Αλλά παρόλα αυτά αυτό που θα έλεγα είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των διάφορων πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει ένα ανοιχτό πνεύμα. Μα καλωσόρισαν ε, τόσο εγκάρδια σε όλη τη διαδικασία. Ήθελαν να είμαστε εκεί θεωρούσαν ότι είναι παραγωγικό ο ρόλο που είχαμε να επιτελέσουμε. Η Επιτροπή σα ε, μιλάει πολύ για τον συντονισμό για του δωρητέ και υποθέτω ότι θα συνεχίσετε να το κάνετε, αλλά μέσω του, το ΟΗΕ και των ε, σχετικών κονδυλίων υπάρχει δυνατότητα συντονισμού δωρητών. Οπότε υπάρχουν αρκετά ε, πλεονεκτήματα ώστε να εγκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα αυτή και αυτό μπορεί όντω να κάνει τη χώρα αυτή λίγο διαφορετική από άλλε. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε τη χώρα αυτή για περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ και εσένα για τα σχόλια που έκανες, ήσουν και σήμερα της αντιπροσωπείας. Είπα και στην παρουσίασή μου στην αρχή, θα το ξαναπώ, σε ό,τι αφορά την Αφρικανική Ένωση, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο μέλλον. Εμείς ήμασταν εκεί περίπου τρει μήνες πριν τι εκλογέ και μπήκαμε πραγματικά ενεργά σε όλη τη διαδικασία. Αλλά οι Αφρικανοί παρατηρητέ αυτό που κάνουν είναι ότι έρχονται την τελευταία στιγμή και δεν το λέω ε, επικριτικά, αλλά ε, επιλέγουν πολύ συγκεκριμένου ε, πολιτικού που είτε έχουν συνταξιδοτηθεί και έρχονται ω παρατηρητέ, αλλά έρχονται τελευταία στιγμή. Ε, αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να είναι πιο έντονη η επικοινωνία μας, να γίνει από πιο νωρί, να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, ίσως και προσωπικά μαζί τους, πριν φτάσουν στη χώρα, για να δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ μας με τους υπόλοιπους Αφρικανούς παρατηρητές και εγώ είμαι περήφανος για αυτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εκλογές ε, και ευχαριστώ και τον Ρικάρντο για τα σχόλιά του. Για τον κύριο Γκέρεν, σε ευχαριστώ που για όσα είπατε. Για την 11η ETF τα είπα. Ε, χρειάζεται η δέσμευση. Χρειάζεται όντω η, θεωρία να γίνει πράξη. Χρειάζεται να υπάρξουν κονδύλια. Ξέρω ότι και ο Επίτροπο Πίμπελξ ασχολείται με το θέμα αυτό. έτσι ώστε να μπορέσουμε να, α, οι καλές μας προθέσεις να μετατραπούν και σε συγκεκριμένες πράξεις. Τώρα, για, την, για τις διάφορες εκστρατείες. μέσω μεγάλων ε, ε, διαδηλώσεων ε, γίνονται αυτές οι εκστρατείες με πολύ δυνατή μουσική, με αλκοόλ, ίσως καμιά φορά και με ναρκωτικά, με χρήματα που αλλάζουν χέρια. Αυτό είναι ο τρόπος που γίνονται οι διάφορες πολιτικές εκστρατείες των, κρατών των πολιτικών κομμάτων. Συγγνώμη. Και αυτό θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ε, Προφανώ κάποιοι έχουν περισσότερα κονδύλια από άλλου, έχουν περισσότερε ευκολίε από άλλου. Εκεί υπάρχει, υπάρχει μια στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η, Οι εφημερίδες εισάγονται στην ε, πρωτεύουσα, στο Freetown και διαβάζονται περίπου από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι λοιπόν αρκετά δύσκολο να υπάρξει να υπάρξουν κάποια πρότυπα αντικειμενικά για, την, ε, ε, για τους δημοσιογράφους και για την ε, καταγραφή των άρθρων τους. Εδώ λοιπόν μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο. Έγινε και μια συζήτηση μεταξύ της δικής μας αντιπροσωπείας και του κρατικού τηλεοπτικού φορέα για το τι χρειάζεται και ήθελα αυτό να, το, σας, το, να σας το πω. Έχουμε δώσει σαφεί ενδείξει εμεί και για τα ΜΜΕ και για το τι μπορεί να γίνει. Έχουμε κάνει κάποιε προτάσει. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά και από τον BBC και από δημοσιογράφου που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε και βεβαίως θα με εκπλήσατε αν λέγατε ότι διαφωνείτε με την ανάλυση που κάναμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπατε 100%. Και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και του δικού σα συναδέλφου, όσου ε, βρίσκονται στι ομάδε που υποστηρίζουν τι ε, αποστολέ των χώρων αυτών εδώ στι Βρυξέλλε. Πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και σα παρακαλώ να μεταφέρετε τι ευχαριστίε μου. Νομίζω ότι όντω ε, ο πρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων έκανε μια σαφή αναφορά στον πολιτικό διάλογο. Υπάρχουν δύο κόμματα στη χώρα αυτή έχει, υπάρχει η ιστορία του εμφυλίου ε, πολέμου, υπάρχει πραγματικά μεγάλη ε, αναξιοπιστία μεταξύ των δύο και είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί ένα έστω ελάχιστο επίπεδο συνεργασίας ε, που είναι κάτι που χρειάζεται για να υπάρχει μια σχέση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Για να δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να δημιουργηθούν και κάποιοι μηχανισμοί. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι του δικού μα έργου από εδώ και μπρο. Η Βερονίκ με ρώτησε για το κατά πόσο είναι έφραυστη η δημοκρατία στη χώρα αυτή. Αυτή νομίζω ότι ήταν η στιγμή όπου η δημοκρατία πραγματικά άρχισε να ισχυροποιείται. Πρέπει να πω όμως ότι ένα υπήρξε ένα σημείο μετά τις εκλογές όπου η, η, αντιπολίτευση δεν τις δέχτηκε, ε, είχε κάποιους ε, οπαδούς της ε, στους δρόμους που ζητούσαν να γίνουν έλεγχοι, που απειλούσαν να μποϊκοτάρουν το κοινοβούλιο και μέσω μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων της, αντιπροσωπ... της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση δεν κατάφερε το πρόβλημα να λυθεί Μάλλον κατάφερε το πρόβλημα να λυθεί, αλλά για να, να εξακολουθήσει να βελτιώνεται η κατάσταση, ε, θα πρέπει να, να υπάρξει υποστήριξη. Ε, ένας από τους δύο πολιτικούς ηγέτες, ε, σε μία από τις πρώτες συναντήσεις του μαζί μας, μας είπε ότι υπάρχουν 90.000 αστυνομικέ δυνάμεις και ειρηνευτικές δυνάμεις εδώ στη χώρα μας. Εγώ έχω 60.000 υποστηρικτές στα βουνά. Αν δεν περάσει αυτό που θέλω στις εκλογές, αυτοί οι 60.000 από τα βουνά θα κατέβουν στο κέντρο και είπε για την κυβέρνηση ότι δεν θα τους στείλω στο Διεθνές Δικαστήριο γιατί θέλω να τους κρεμάσω εγώ πρώτα. Και αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές που λες τι απαντάει κανείς. Εγώ απλώ τον κοίταξα και του είπα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει την ποινή του θανάτου αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούσα να του δώσω εκείνη τη στιγμή. Αλλά οι δικέ του απειλέ βεβαίω ε, ήταν κενέ. Ε, Προφανώ το ε, κόμμα του δεν έτυχε μεγάλη υποστήριξη και αυτό είναι και ένα από τα, από τα μηνύματα που πρέπει να εξάγουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί η δημοκρατία σε χώρες όπως η Σιέρα Λεόνε. Η Ευρώπη λοιπόν μέσω της αποστολής της ε, πρέπει να το παρακολουθεί και γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα στις χώρες αυτές και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη χώρα αυτή που είναι μια πανέμορφη χώρα και που μας ε, καλωσόρεσε πραγματικά εγκάρδια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Χάουιτ, πολύ σημαντική η εμπειρία σας από τη Σιέρα Λεόνη και σας ευχαριστούμε που τη μοιραστήκατε μαζί μας. Πάμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα αναπτυσσόμενα κράτη. Θα γίνει μια παρουσίαση μιας μελέτης. Την αναθέσαμε αυτή τη μελέτη. Προετοιμάστηκε από το Οικολογικό Ινστιτούτο που εξετάζει την βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η μελέτη διεξήχθη από την κυρία Φραντσέσκα Παστάλια, που είναι παρούσα, είναι εδώ μαζί μας, και στην οποία δίνω αμέσω το λόγο για να μας παρουσιάσει τα βασικά πορίσματα της εκθέσεως. Η κυρία Μπαστάλιο λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα για να σας παρουσιάσω τα βασικά συνοπτικά πορίσματα τη εκθέσεω που μα ανετέθη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέποντα πόσο είναι εφικτά τα συστήματα κοινωνική προστασία στα αναπτυσσόμενα κράτη. Θα ακολουθήσω το πλαίσιο που μου ετέθη. Η παρουσίαση αυτή κοινά του στόχου για την κοινωνική προστασία, τα εργαλεία, εστιάζεται επί θεμάτων κάλυψη και τι γίνεται στις χώρες που είναι λιγότερο εντυγμένες με χαμηλό εισόδημα πώς προωθείται η κοινωνική ασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες, ποιος είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και στο τέλος θα αναφερθούμε στις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά ε, το διεθνές ε, πεδίο για την προώθηση της κοινωνικής προστασίας και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Το ιστορικό. Πρέπει να τονίσουμε ότι η κοινωνική προστασία έχει πολλαπλούς στόχους η παρουσίαση αυτή εστιαζόταν συγκεκριμένα στην κάλυψη ε, και τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας έχουν και άλλους στόχους. Ένας από αυτούς είναι η εξομάλυνση του εισοδήματο και της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της ζωής, ώστε τα άτομα και τα νοικοκυριά βοηθούνται για να αντιμετωπίσουν διαφόρους κινδύνους κατά τη διάρκεια της ζωής, ανεξάρτητα από το εισόδημά του ότι είναι χαμηλού εισόδηματο νοικοκυριά. Άλλα προγράμματα κοινωνική προστασία έχουν στόχο σαφή τη μειώσεως τη ένδυα. Άλλοι στόχοι είναι η ανακατανομή σε άλλα προγράμματα. Και πρέπει να τονίσω ότι η μείωση τη ένδυα και η μείωση των ανισοτήτων δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα. Ένδια και ανισότητα έχουν κάποια αλληλεπικάλυψη, αλλά είναι διαφορετικά θέματα και διαφορετικά αποτελέσματα. Άλλη διάκριση πρέπει να κάνουμε είναι μεταξύ προγραμμάτων κοινωνική αρρωγή και προγραμμάτων κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική βοήθεια, κοινωνική αρρωγή είναι κάτι που χρηματοδοτείται από τον φόρο, από τη φορολόγηση και αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά και ευάλωτε ομάδε. Η κοινωνική ασφάλιση, από την άλλη, εν γέννη χρηματοδοτείται μέσω εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών και αφορά ανθρώπους που εργάστηκαν κάποιους ή έχουν όριμα δικαιώματα και κοινωνική προστασία μέσω της πρώτερης ε, απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας. Και τέλος, δεν υπάρχει συμπεφωνημένος ορισμός για την κοινωνική προστασία, άρα συζητείτε και είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καμιά φορά περιπλέκονται οι συζητήσεις λόγω της ελλείψης ορισμού. Υπάρχει φάσμα ορισμών, δεν θα αναφερθώ σε όλους τους ορισμούς, ποικίλουν από μινιμαλιστική προσέγγιση όσον αφορά τις παρεμβάσεις, δίκτυα ασφαλείας, που τα δίκτυα ασφαλείας προσπαθούν να καλύψουν τα νοικοκυριά και τα άτομα που δεν καλύπτονται από τα συστήματα, τα δημόσια και από τις αγορές, το άλλο άκρο. Διάφορες παρεμβάσεις που προσπαθούν εν γέννη να προωθήσουν την ευημερία δεν είναι μόνο στοχευμένες παρεμβάσεις, αλλά γενικά προγράμματα που προστατεύουν, προωθούν και μετατρέπουν, αλλάζουν την ευημερία των πολιτών. Τώρα, υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα ε, όσον αφορά προστασία. Ε, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες μεταφορές σε μετρητά, σε είδος, φορολογικά και χρηματοπιστωτικά μέσα ελαφρύνσεις φορολογικές παραδείγματος χάρη και εξαιρέσει και διάφορα προγράμματα δημοσίων έργων και δραστήριες ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και από τις γενικές κατηγορίες έχουμε υποκατηγορίες μεταφορές και εμβάσματα σε ρευστό ε, μπορούν να τελούν υπό προϋποθέσεις όταν οι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθούν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι και ανεφόρων η παροχή των ε, χρημάτων ε, πολύ συχνά οι συζητήσεις θεάζονται επί του ποια, ποιες είναι βέλτιστες και προτιμητές. Δυστυχώς λέγω διότι το επιθυμητό μιας επιλογής σε σχέση με άλλη εξαρτάται από τον επιδιωκόμενο στόχο και από τις περιστάσεις τις συγκεκριμένες ε, για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται μια πολιτική ποιοι είναι οι λόγοι για χαμηλή κάλυψη όσον αφορά την κοινωνική προστασία σε χώρες με χαμηλό εισόδημα. Έχουμε τρεις λόγους βασικούς. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη χρηματοδότηση, πόρους. Δεύτερο, οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού πολιτικών και εφαρμογή των πολιτικών. Και τρίτη πτυχή, πολιτική οικονομία και διάφορες τέτοιες πτυχές. Επίπεδα χρηματοδότησης. Τα επίπεδα, όπως φαντάζεστε και όπως γνωρίζουν πολύ καλά, ε, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι σε χώρες με υψηλό εισόδημα ή μεσαίο εισόδημα και αυτό εξηγεί εν μέρη και το χαμηλό αποτέλεσμα ή αμελητέ αποτέλεσμα που διαπιστώνεται όσον αφορά την ένδια και την ανισότητα σε χώρες με υψηλό εισόδημα όπου σημαντικά ποσά των δημοσίων δαπανών αφορούν ε, την κοινωνική προστασία και τις σχετικές δαπάνες υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος όσον αφορά την ανισότητα των εισοδημάτων και όσον αφορά άλλε ανισότητες πέρα από το επίπεδο των δαπανών υπάρχει και το θέμα του μείγματο των δαπανών. Από πού προέρχονται τα χρήματα. Και υπάρχει σαφής διάκριση των όσων συμβαίνουν στι χώρε με χαμηλό εισόδημα σε συγκρίση με τι χώρε με ψηλό εισόδημα. Είναι και το εξή. Μεγάλο ποσοστό των πόρων τη χρηματοδοτήσεω προέρχεται από οικονομίε νοικοκυριών, ιδιωτικέ δαπάνε κλπ. Και δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η κοινωνική προστασία χρηματοδοτείται κατά πολύ από εξωτερική βοήθεια. Ε, και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έχουν διάφορες ε, συνέπειες που θα αναφέρουμε αργότερα, αλλά εν συντομία εδώ θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι πληρωμές από τον ιδιωτικό, από αποθέματα, από την τσέπη ε, περιορίζουν σημαντικά την κατανάλωση και το εισόδημα των φτωχών οικοκυριών. Ε, δεύτερη πηγή χρηματοδότησης για την κοινωνική προστασία στις στοχές χώρες είναι η εξωτερική βοήθεια και οι δωρητέ. Άρα εκεί αμφισβητεί την νομιμότητα των προγραμμάτων και κατά πόσον έχουν συνέχεια τα εφαρμοζόμενα προγράμματα. Πάμε τώρα σε άλλε λεπτομέρειε. Αν σκεφτούμε τις λεπτομέρειες της κοινωνικής ε, βοήθειας, ε, προφανώς ε, εξορισμού καλύπτεται το πώς σχεδιάζονται όλα αυτά τα προγράμματα, ε, ποιους στοχεύουν, ποιες, υπό ποιες προϋποθέσεις δίνονται. Τα προγράμματα αυτά περιορίζονται σε πολύ μικρό ποσοστό αυτού του, ε, ε, του πληθυσμού και βεβαίως αυτό προφανώς περιορίζει και την κάλυψη. Όπως έχει γράψει και ο Τόνι Ακκινσόν, ο στόχος θα μπορούσε να οριστεί σε πολλές χώρες διαφορετικά. Για πολλές χώρες ακόμα οι στοχοθέτηση είναι πολύ περιορισμένοι. Για τα προγράμματα που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση, ε, ένα, ένα μία από τις βασικές προκλήσεις είναι ε, το άτυπο ε, σύστημα που υπάρχει σε πολλές χώρες και βεβαίως η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει άτομα που πληρώνουν τις κοινωνικές τους εισφορές. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εξαιρείται από, τέτοιες, από τέτοια προγράμματα κοινωνική ε, πρόνοια. Και αν δούμε και τις λατινοαμερικανικές χώρες, ε, τα προγράμματα τα μέχρι πρόσφατα ε, αποτελούνται ουσιαστικά από κάποιους διακανονισμούς με την άτυπη η οικονομία και αυτό βεβαίως οδήγησε σε ένα εντελώς κατακαιρματισμένο σύστημα, ένα μεγάλο δηλαδή κομμάτι του εργαζόμενου πληθυσμού δεν καλύπτεται από την κοινωνική πρόνοια. Αυτό τα τελευταία χρόνια ε, προσπάθ, έγιναν προσπάθειες να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μέσω εμβασμάτων έτσι ώστε να μπορέσει να καλυφθεί περισσότερο κομμάτι των χαμηλών εισοδημάτων και των εργαζομένων. Τώρα πάμε στις ε, διάφορες ε, λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα αυτά. Το, αποτέλεσμα, ε, το, το πρόβλημα μάλλον προκύπτει από ε, την απουσία συμφωνίας, πολιτικής συμφωνίας ή κοινή συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το ποιοι θεωρούνται ευάλωτοι και ποιο είδος κοινωνικής προστασίας ε, τους, πρέπει να τους παρασχεθεί. Αν δούμε λοιπόν τις, ομάδες που έχουν, τις χώρες που έχουν καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού τους με κοινωνική προστασία, αυτές οι χώρες το κατάφεραν επειδή έχει υπάρξει κάποιο είδος κοινωνικού συμβολέου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική προπόθεση για να μπορέσει να διευρυνθεί η κοινωνική προστασία και ε, πάει χέρι-χέρι με την ε, βελτίωση και την προώθηση ε, της εκπροσώπησης των ομάδων που συνήθω δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα συστήματα κοινωνική πρόνοια. Μία δεύτερη λεπτομέρεια έχει να κάνει με, την, το σχεδιασμό τη πολιτική και όπω ξέρουμε και μα μας το λέει και η βιβλιογραφία τα προγράμματα αυτά που περιλαμβάνουν πολύ μικρό πληθυσμό προφανώς δεν υποστηρίζονται και από τον πληθυσμό. Και όπως ε, έχει αναφερθεί εδώ και πολλά χρόνια, η πολιτική για τους φτωχούς είναι φτωχή πολιτική. Πάμε τώρα στην κοινωνική ασφάλιση. Ένα από τα προαπαιτούμενα είχαμε πει ότι θα συζητούσαμε το πώς θα μπορούσε να διευρυνθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι που το, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν να ε, επεκταθούν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Ήδη σας μίλησα για τις, ε, για τις μικρές επίσημες οικονομίες και την μικρή συμμετοχή στην επίσημη οικονομία που προφανώς διακυβεύει την συμμετοχή και την διεύρυνση της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, ε, τα είδη του κινδύνου που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα Επίσης υπάρχει έξτρα κόστος που σχετίζεται με την ε, ε, ασφάλιση των ε, χαμηλών εισοδημάτων και αυτό έχει να κάνει και με την ενημέρωση και με τη δυσκολία λήψης πληροφοριών ώστε να μπορέσει να διευρυνθεί το πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης και το θέμα είναι και η περιπλοκότητα και, το, και τα προσόντα που έχει ένας άνθρωπος χαμηλού εισοδήματος ε, και το πώς μπορεί, πόσο μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς δικαιούται. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται λεπτομερέστερα με παραδείγματα στην ε, σχετική ενημέρωση. Τώρα, η τυποποίηση μπορεί να προωθηθεί, μπορεί να βελτιωθεί με, αρκετό, με αρκετούς τρόπους. Ένας από αυτού είναι να βελτιωθεί η κατάρτιση σε όσους βρίσκονται στην άτυπη αγορά, να ενημερωθούν καλύτερα οι εργαζόμενοι, να, πληροφορηθούν, να τους δοθούν περισσότερε πληροφορίε, να κλείσουν τα κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση, να μειωθούν οι ανισορροπίε, οι ανισότητες που υπάρχουν. Επίση πρέπει να προωθηθεί έτσι ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι εργαζόμενοι που μπαίνουν ή βγαίνουν από την αγορά εργασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να του ενθαρρύνουμε να ε, συμμετέχουν ε, στην επίσημη ε, οικονομία και στα επίσημα προγράμματα κοινωνική ασφάλισης. Αυτό είναι μια σημαντική επιλογή που έχουμε. Πέραν αυτού, έχει υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά την παροχή κοινωνικής ασφάλισης. Νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό να είμαστε σαφείς. Υπάρχουν διάφοροι παίκτε. Ε, υπάρχει η κυβέρνηση βεβαίω, υπάρχουν οι, ε, οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, υπάρχουν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αλλά υπάρχουν και εκτός αυτών άλλες ομάδες ε, και άλλοι μπλεκόμενοι φορείς που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε διάφορα επίπεδα εξουσίας και θα μπορούσαν όντως να συμμετάσχουν ή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιε ενώσει ε, κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών ε, οργανισμών. Έχουν λοιπόν διαφορετικέ διαφορετικές σε κάθε ομάδα. Μιλούμε για ε, έλεγχο, μιλούμε για εποπτεία, μιλούμε για χρηματοδότηση της κοινωνική ασφάλισης και μιλούμε και για την παροχή αυτή καθ' αυτή της κοινωνική ασφάλιση. Η ενημέρωση παρέχει κάποια παραδείγματα για τις διάφορες οργανώσεις ε, και το πώς αυτές μπορούν να συμβάλλουν στις διάφορες λειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης. Αλλά αν κάνουμε ένα βήμα πιο πίσω και δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κοινωνική ασφάλιση, θα δούμε ότι ο ιδιωτικός τομέας ε, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, η συμμετοχή του δηλαδή, μπορεί να βελτιώσει την ευελιξία των ε, συστημάτων ε, και της παροχής οικονομικής ασφάλισης μπορεί να δώσει μεγαλύτερη επιλογή. Στη θεωρία όλα αυτά μπορούν να συμβούν. Στην πράξη λίγες είναι οι αποδείξεις στα πλαίσια του ΩΣΑ τουλάχιστον ότι αυτό έχει όντω γίνει. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η, ε, η πλήρης ιδιωτικοποίηση μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες ανησυχίες. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη η θεωρία είναι καλή, αλλά θα πρέπει να δούμε και στην πράξη πώ ε, μεταφράζονται όλα αυτά. Αν θέλουμε τώρα να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε περιπτώσει όπου η συμμετοχή των ε, κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών έχει όντως βοηθήσει για να φτάσει η κοινωνική ασφάλιση σε κάποιες ομάδες ε, πολιτών που μέχρι τότε εξαιρούνται. Ας πούμε, η τα, ε, τα κοινοτικά προγράμματα κοινωνικής ή ιατρικής ασφάλισης που υπάρχουν σε πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αυτά είναι προγράμματα που είναι τοπικά και που τυπικά γίνονται, ε, ε, εξελίσσονται μέσω πληρωμών σε ένα ταμείο. Η κοινότητα παίζει σημαντικό ρόλο βεβαίως στο να αποφασίσει πώς θα διανεμηθούν αυτά τα κονδύλια αυτό είναι το σύνηθε ε, σε, τέτοιες, ε, σε τέτοια προγράμματα κοινωνική ασφάλιση τοπικά. Και αυτό που βλέπουμε σε πολλέ χώρε, όπω σε Σενεγάλη ή σε χώρε στην Ινδία, είναι ότι ε, αυτά τα προγράμματα τα τοπικά όντως έχουν συμπεριλάβει πολλές ομάδες χαμηλού εισοδήματο που μέχρι τότε δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να καλύψουν τα ιατρικά τους έξοδα. Οπότε αυτό είναι αρκετά σημαντικό ως αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα έχουμε δει ότι υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι οι πιο φτωχοί εξακολουθούν να εξαιρούνται. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων η μόνιμη, ο μόνιμος αυτός αποκλεισμός προκύπτει από την ανικανότητα των ομάδων με χαμηλό εισόδημα να συμβάλλουν σε αυτή την προπληρωμή έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτά τα τοπικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης. Άλλοι λόγοι εξαίρεσης έχουν να κάνουν με τον τόπο που, που ζουν, δηλαδή ε, περιοχές που δεν καλύπτονται, που δεν υπάρχουν καταστάσεις και δεν μπορούν να συμμετέχουν ω περιοχές σε, σε αυτά τα προγράμματα. Και επίσης, ο ρόλος της κυβέρνησης που σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχει περιθώριο παρέμβασης ε, μη κερδοσκοπικών, ιδιωτικών ή κερδοσκοπικών οργανισμών να προωθήσουν την ασφάλιση, η κυβέρνηση εξακολουθεί να παρεμβαίνει και να προωθεί την συμμετοχή, εξασφαλίζοντας ότι θα διευκολυνθεί αυτή ακόμη και για τους πολύ πολύ φτωχούς ας πούμε μέσω ε, κάποιων ε, ε, ελαφρύνσεων φορολογικών για ανθρώπους με πολύ χαμηλό εισόδημα έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν κάποιο μέρος των πληρωμών αυτών ή επίσης φροντίζοντας να υπάρχουν καταστάσεις σε όλη τη χώρα, στην επικράτεια της χώρας και η ποιότητα των καταστάσεων αυτών θα είναι ενό επίπεδου αξιόπιστου για να μπορούν ε, να στρέφονται σε αυτές οι ακόμη και οι πιο φτωχοί. Προχωρούμε. Γίνεται μια αναφορά στην ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις ε, σε διεθνές επίπεδο, για τις ε, Προσπάθεια προώθησης τη ε, κοινωνική ασφάλισης, του συντονισμού διαφόρων ε, πρωτοβουλειών για την κοινωνική ασφάλιση. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι θα ξέρετε το Social Protection Floor του ILO που έχει ξεκινήσει ε, εδώ και δύο χρόνια και που έχει αναγνωριστεί από πολλέ οργανώσει. Η G20 επίση το έχει αναγνωρίσει και άλλοι οργανισμοί, οι υπηρεσίε του ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα επίση, όλοι συνεργάζονται ε, με τον ILO για την προώθηση των ε, εθνικών ε, προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό φαίνεται ότι υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κοινωνική ασφάλιση μετά και την οικονομική κρίση και το ότι φαίνεται και από τις επενδύσεις στην κοινωνική ασφάλιση. Και οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές και για το μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ευημερία των πολιτών και στο μέλλον και σε σχέση με μελλοντικέ κρίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, ποιο είναι ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα, πολύ, ένα μοναδικό εργαλείο, είναι η μοναδική θέση που έχουμε και λόγω της σταθερής παράδοσης που έχουμε στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, παρά τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στην, στα διάφορα κρατημέλη, εξακολουθεί να υπάρχει μακρά παράδοση ε, παροχής κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη και τη δυνατότητα να προωθήσει τέτοιου είδους ε, προγράμματα και σε χώρες χαμηλού εισοδήματο. Ε, υπάρχουν τρία είδη δράσεων, όπως η υποστήριξη άμεσα ε, των κυβερνήσεων για την χάραξη τη πολιτικής και την εφαρμογή, τη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλειών, η προώθηση της ε, ενημέρωσης και της κατάρτισης, καθώς επίσης και η ε, αξιολόγηση και η εποπτεία. Και ένα τελευταίο πίνακα θα δείτε εδώ, που υπάρχει και στην ενημέρωση, όπου παρέχονται παραδείγματα για τους, με, από, τη μια, με, ε, των περιορισμών που υπάρχουν στην παροχή κοινωνική κοινωνικής ασφάλισης, όπως η χρηματοδότηση, όπως η χαράξη πολιτικής, όπως η οικονομία και καταγράφονται και κάποιοι τομείς που θα μπορούσαν να υπάρξει στήριξη. Δράσεις δηλαδή που θα μπορούσαν ε, να ε, υπάρξουν μέσω της ε, αναπτυξιακής βοήθειας, αναπτυξιακής συνεργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, madame. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ντικεζέρη, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία για την παρουσίαση. Είναι γεγονός ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό, δηλαδή της κοινωνικής ε, ασφάλισης και προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, αλλά ξέρετε κάπως... Ε, έχω μπερδευτεί. Εμείς εδώ συντάξαμε μια έκθεση εγώ ήμουν σε τραβέβα, αλλά πήρα ε, υπόψη μου τα σχόλια όλων των συναδέλφων για το ίδιο θέμα, στην αρχή τη θητεία. Και θυμάμαι πολύ καλά κάποιε από τι ε, διαπιστώσει έκθεση. Η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι σχεδόν καμία αναπτυσσόμενη χώρα δεν μπορεί με τον προπολογισμό που έχει να εξασφαλίσει στην κυβέρνηση τους απαραίτητους πόρους για να καλύψει τις δαπάνε αυτές, άρα θα πρέπει να υπάρχουν εξωτερικοί πόροι που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν σε μια κυβέρνηση τις απαραίτητες υποδομές ε, για την υγεία, ε, για το ιατρικό προσωπικό και ούτω καθεξής. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι κάπου να δώσουν τις εισφορές τους για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές τις εισφορές για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας λοιπά, Για τους πιο φτωχούς. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα οποία έχω δει και έχω ακούσει μπορώ να τα πιστέψω. Δεν θα ήταν καλό να υπάρχει ε, μια κουλτούρα ε, τέτοια στις περισσότερες χώρες και εσείς σε αυτό που είπατε community base περιγράφεται. Περιγράφεται ότι υπάρχουν αυθόρματα κάποιες μικρές δομές αλληλοβοήθειας που θα πρέπει να ενισχυθούν. Τι στηρίζουν κάποιες φορές ε, οι ενορίες, για παράδειγμα, οι μη κυβερνικέ οργανώσεις. Είναι λοιπόν κάποιες δομές αλληλεγγύης. Υπάρχουν και πρέπει να τις ενισχύσουμε απλά, να τις κάνουμε να εξαπλωθούν. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω χιλιάδες τέτοιες δομές. Όμως υπάρχει μια τεράστια αγορά για τον ιδιωτικό τομέα για τις πιο πλούσιες όμως κατηγορίες του πληθυσμού. Γιατί λέω ότι με μπέρδεψε η παρουσίασή σας, με αποπροσανατόλισε, διότι όταν μιλάμε για το δυνητικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στο περιβάλλον της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί μιλάμε ακριβώς, τι εννοούμε, ποιον ιδιωτικό τομέα Μιλάμε για αυτές ε, τις ε, τους συντερισμούς ενδεχομένως ή τις εταιρείες αλληλασφάλισης. Εγώ στο Βέλγιο ξέρω ότι υπάρχουν ε, οργανώσεις που ενισχύουν, ε, παραδείγματο χάρη, οργανώσεις ε, στην Πασαχάριο Αφρική. Ακριβώς αν θέλετε για να μην είναι οι, οι υπηρεσίες αυτές στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, να μην μπαίνουν δηλαδή τα λεφτά στις τσέπες κάποιων ε, γιατί μιλάμε λοιπόν ακριβώς τελικά. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτό που είπαμε εμεί στη δική μα έκθεση και αυτό που μα περιγράφετε εσεί και δεν λέω ήταν αυτή η έκθεση αχρίαστη σε καμία περίπτωση, αλλά για ποιον ιδιωτικό τομέα μιλάμε και τι πιστεύετε για του πιο φτωχού. Μήπω ακριβώ το αντίθετο θα πρέπει να συμβαίνει, όχι μέσω ιδιωτικού τομέα, αλλά να στηρίξουμε την τοπική αλληλεγγύη, τι τοπικές δομές αλληλεγγύης. Η Πρόεδρος δίνω το λόγο σαν εαυτό μου τώρα. Και εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την παρουσία της κυρίας Φραντσέσκα Παστάλη και πρέπει να πω ότι και μένα με ξένησε η πολύ αφηρημένη ε, παρουσίαση ουσιαστικά. Εγώ θα ήθελα να έχω συγκεκριμένα παραδείγματα να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα συστημάτων που κατάφεραν να καλύψουν ένα τμήμα του πληθυσμού ή να δούμε και παραδείγματα τα οποία αντιθέτω έδειξαν ότι δεν ε, απέδωσαν. Νομίζω ότι λείπουν ε, τα νούμερα, τα πραγματικά στοιχεία, τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Και όταν λέτε ότι υπάρχει για τον ιδιωτικό τομέα πολλής χώρος, τι εννοείται ακριβώ. Παραδείγματο χάρη, στη Μοζαμβίκη οι εταιρείε, οι εξορρυκτικέ που δεν πληρώνουν φόρο, εξασφαλίζουν την κοινωνική προστασία των εργαζομένων του που μοιάζουν με σκλάβοι ουσιαστικά. Πολύ θα ήθελα να μου πείτε πάνω σε αυτό κάτι. Επίση, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον σε αυτές τις μελέτες υπολογίζεται με τον ένα τον άλλο τρόπο οι πόροι που δεν έχουν ε, τα κράτη και με τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις υπηρεσίες μέσω κάποιων παράνομων ε, μεθόδων και κυκλωμάτων. Παραδείγματο χάρη δεν υπάρχουν, ε, δεν, δεν εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση στις χώρες αυτές παραδείγματο χάρη τα έσοδα από δασμού ή τέτοια, παραδείγματα. Αυτά θα ήθελα να ακούσω από εσά. Ο κύριο Μίτσελ τώρα, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, στο συγγνώμη που άργησα το θέμα αυτό έχει μπει στην μέση διάταξη γιατί το ζήτησα εγώ, ίσω και άλλοι βέβαια φαντάζομαι, αλλά και γιατί είχα ζητήσει να το βάλουμε στην μέση διάταξη, κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ άλλων, γιατί πίστευα ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε πάρα πολύ ε, στα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, στον ανυψόμενο κόσμο, λίγο πολύ ε, ε, όλοι είναι φιλόδεξος εμείς, τα παιδιά είναι ικανά ως τα δικά μας αλλά είναι πολύ άριθμες οικογένειες εκεί, κυρίως διότι πιστεύουν ότι αυτό θα τους δώσει ασφάλεια για το μέλλον και δεν μπορούν να τη βρουν αλλιώς αυτή την ασφάλεια, άρα πολλά παιδιά γεννάνε γιατί πιστεύουν ε, ότι θα τους παράχουν αυτά. Και βέβαια σίγουρα αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και για τις οικογένειες, για τις μητέρες, ε, για το ιατρικό σύστημα, για πολλά και διάφορα. Αν δείτε όμως το δικό μας μοντέλο, εδώ όλοι μας. Όλοι θέλουμε κοινωνική ασφάλιση και προστασία. Αν αρρωστήσουμε, αν είμαστε στη σύνταξη, αν έχουμε άδεια μητρότητα, πατρότητα και το καθεξής. Άρα, αυτό που να σας ρωτήσω είναι, πρώτον, έχουμε νομική βάση. Το DCI το καλύπτει από ό,τι κατάλαβα. Τι δεν καλύπτεται, ό,τι δεν καλύπτεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε κάποια δυνατότητα νομική να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρήματα για να τα προωθήσουμε. Και εμείς ως βουλευτές θα μπορούσαμε να κάνουμε για να κινηθούν κάπως τα πράγματα. Πού πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για να ε, κινηθεί λίγο το πράγμα. Και τρίτον, η Κομισιόν πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον να δράσει ως καταλήτης δηλαδή να επιλέξετε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ίσως και μια πιλωτική περιοχή, μια πιλωτική χώρα, ώστε να μας πείτε πώς θα μπορούσε να έχει καταλυτικό, καταλυτική δράση κομισιών. Ε, δεν ξέρω τι εννοούμε τώρα, ένα μοντέλο ε, ε του, ένα μοντέλο ιδιωτικού τομέα. Τι μπορούμε να δοκιμάσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να παράσχουμε κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική προστασία στον κόσμο για να μην νομίζει ότι έχει μόνο ε, μία διέξοδο, δηλαδή να γεννήσει πολλά παιδιά. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ο πυρήνα των προβλημάτων, γιατί ο κόσμος εκεί δεν έχει εναλλακτικέ. δεν νιώθει να έχει εναλλακτικέ. Θα το εκτιμούσα λοιπόν να μας δίνετε τις απόψεις Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίαση, αλλά επειδή άρχισε η πτήση μου, ζητώ συγγνώμη που έχασα την αρχή της παρουσίασης. Κύριος Μαρτίνες, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με τη σύγχυση που την επετελεί η κυρία Τεκάιζερ. Συμμερίζομαι και τα δικά σας σχόλια, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ έτσι θα αντιδρούσα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Αν μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση και προστασία, ουσιαστικά μιλάμε προστασία της κοινωνικής ασφάλισης. Από τότε που γεννάται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει ένας πολίτης μιας χώρας. Από ενολική πλευρά, επομένω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφορά σε αυτό μεταξύ αναπτυγμένων, αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ φτωχών και πλούσιων. κάθε πολίτης από οποιαδήποτε χώρα έχει ως θεμελιώδης δικαίωμα την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει. Γι' αυτό μιλάμε. Και αυτή η κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνει υγεία, σύνταξη, Είτε μιλάμε βέβαια ε, για επίδομα ανεργίας, είτε μιλάμε για σύνταξη αυτή καθεαυτή. Επιδόματα δηλαδή τελικά. Εσείς έχετε περιλάβει την παιδεία, δεν ξέρω ε, αν την συμπεριλαμβάνετε σε αυτούς τους τομείς, στους οποίους η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να ισχύει και να εφαρμόζεται. Επίσης, Το λέτε στην έκθεσή σας, αλλά κάπως ε, μέσα σε κάποιες άλλες ιδέες ψιλοχάνεται, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε ως χαρακτηριστικό τη γενίκευση της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης ως δημόσια ευθύνη. Ανεξαρτήτως δηλαδή το αν ένας πολίτης είναι νέος, γέρος, ε, φτωχός, πλούσιος, αν ζει στη θάλασσα, αν ζει στο βουνό. Έχουμε μια καθολική δημόσια ευθύνη για την παροστασία της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προβάλλουμε όχι μόνο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά να θεωρήσουμε ότι είναι και θεμητή προσδοκία και φιλοδοξία των ανδρών και των γυναικών που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε αναπτυσσόμενο κόσμο. Ε, Επομένω, αυτό που μου φαίνεται προφανέ είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που έχουμε τελείως διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις. Αυτή λοιπόν η ανάληψη ευθύνη, η υπευθυνότητα του δημόσιου τομέα, του κράτου για μα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια συνυπάρχει και με το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό και γενικότερα με τις δράσεις μας, αλλά και σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση και την κρίση που βιώνουμε και που βλέπουμε κάποιες από αυτές τις πτυχές που θεωρούσαμε τα χαρακτηριστικές με κάποια αφέλεια θεωρούσαμε ότι είναι και αμετάκλητες, ε, βλέπουμε ότι υπονομεύονται εδώ. Τώρα, σε αναπτυσσόμενες χώρες, επειδή είναι άλλες οι ιδεολογικές τοποθετήσεις, γενικεύεται και εκεί η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης. Σε μια χώρα όπως η Κούβα, η ουσία του κουβανικού κράτου. Μπορεί να κανεί να συμφωνεί ή να μην συμφωνεί, αλλά είναι ακριβώ η απόλυτη προστασία τη κοινωνική ασφάλεια. Αυτή είναι η πεπτουσία σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία και τα επιδόματα. Συντάξει ή επιδόματα ανεργία. Στην Ισπανία έχουμε τη λεγόμενη εξάρτηση. Τι θα πει αυτό. Δηλαδή ότι δεν καλύπτεται αλλά που θα πρέπει να είναι φιλοδοξία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι και χρειάζονται μία προστασία, την οποία μπορεί να τους παράσχει οικογένεια, ειδικό προσωπικό, αλλά μόνο βέβαια μπορεί να τους παρασχεθούν αυτές οι υπηρεσίες και αυτή η φροντίδα εάν χρηματοδοτείται από τις δημόσιες κρατικές αρχές Κάτι τώρα που λείπει, δεν το άκουσα από την παρουσίασή σας δεν ήθελα να μου πείτε. Η συνεργασία, η ευρωπαϊκή συνεργασία πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει ως στόχο οι πολίτες των αψόμενων χωρών να μπορούν να απολαμβάνουν αυτή τη δημόσια προστασία της κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχει όμως και η λεγόμενη τριγωνική συνεργασία για τέτοιες δραστηριότητες που λειτουργεί πολύ καλά σε ορισμένες χώρες του κόσμου, όπως στην Αφρική. Δυστυχώ όμως δεν συμβαίνει αυτό όπω εμεί θα θέλουμε μεταξύ Κούβας, ε, Αφρικανικών χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι μεν ε, στην Καραϊβική. Η Κούβα δίνει προσωπικό και γνώση με τη Βενεζουέλα που δίνει πόρους και με τις χώρες με τις οποίες υπάρχει συνεργασία εδάφη, κόπεδα για την ε, ανέγερση νοσοκομείων κτλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεση σας πάντως, είναι ενδιαφέρουσα, αλλά είναι προφανές ότι όπως νομίζω ότι είπε και η κυρία Πρόεδρος, ε, είναι μια έκθεση, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι το πρόβλημα ότι είναι τόσο ουδέτερη ή τόσο αφηρημένη. Πράγματι όμως θα μπορούσε να χαθεί η ουσία τελικά, το συγκεκριμένο. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και αν ε, μιλάμε απλά για κάποιες έννοιες, εντάξει μπορούμε να συμφωνήσουμε πολλά, αλλά αν το διαβιβάσουμε στις χώρες αυτές με τις οποίες έχουμε εταιρική σχέση, ε, ίσως τις ε, μπερδέψουμε και αυτές. Είπε και η Βερονίκ. Μήπως πράγματι υπάρχει ε, αυτό το να έχει κανείς εμπορικό κέρδος, να κάνει, επιχειρή, να κάνει επιχείρηση. Είναι ανήθικο σε κάποιους τομείς. αυτή η προστασία να γίνει μια δραστηριότητα επικερδής. Σας ευχαριστώ. Κόρτες Λάστρα. Πάρα πολύ σύντομα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με τη Βερονίκη με τον Μιχελάνχελ και με την πρόεδρο. Διότι επί της ουσίας, τι είναι διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις άλλες χώρες. Είναι το κοινωνικό τους μοντέλο παρά την κρίση που βιώνουμε. Μια γενική παρατήρηση όμως θέλω να κάνω. Και η έκθεση που μας παρουσιάσατε έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο πηγαίνει στο κέντρο, στην καρδιά της αναπτυξικής συνεργασίας και στο μέλλον αυτής και στο μέλλον της αναπτυξικής συνεργασίας επαναλαμβάνω. Τι βλέπουμε σε αυτή την κρίση. Και ίσως δεν το έχουμε συζητήσει σε βάθος στην Επιτροπή μας ακόμη. Βλέπουμε επίθεση κατά της αναπτυξικής συνεργασίας. Εσείς εδώ ήρθατε να μας μιλήσετε τη συνεργασία, για τους ειδικούς ε, παράγοντες, φορές λοιπά. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την λεγόμενη ολοκληρωμένη προσέγγιση, η συνεργασία αναπτυξιακή για το μέλλον και λοιπά. Και βλέπουμε και μια σημαντική αλλαγή, ε, τουλάχιστον σε μια αναγνωρίζοντα πενταετίας της κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης, και ίσως δεν έχουμε ακόμη ασχοληθεί επαρκώς. Είναι καλό λοιπόν αυτή η έκθεση να μας κάνει να σκεφτούμε. Θέλουμε να στηρίξουμε την αναπτυξή συνεργασία, τη διεθνή συνεργασία. Αλλά πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον όρο συνεργασία, γιατί ναι, μην είχαμε τα, καλά αποτελέσματα είχαμε αυτό στο CISHIELD μέχρι το 2015, αλλά μπορεί λόγω ε, της κρίσης που θα έχει χτυπήσει ε, να έχουμε πολύ χειρότερα στοιχεία για πιο μετά. Πρέπει να βρεθούν και νέοι πρωταγωνιστές. Αλλά βλέπουμε επίσης και πολλοί να προσπαθούν να κατευθύνουν προς νέους τομείς ε, την αναπτυξική συνεργασία. Και όχι μόνο αυτό, έχω να πω και κάτι ακόμα. Όπως σας είπα, μας διαφοροποιεί από τον άλλο κόσμο το κοινωνικό μας μοντέλο. Αυτό που είναι σαφές είναι Όσο διατηρεί η Ευρώπη αυτό το κοινωνικό μοντέλο, άλλες χώρες μεσής οδήματος θα μπορούσαν να, να υιοθετήσουν, αν τους φαίνεται χρήσιμο και ενδιαφέρον το ίδιο μοντέλο. Εν καιρό κρίση, είπαμε ότι το μοντέλο αυτό έχει πληγεί. Θα πρέπει να δούμε ίσως ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο για να αναπτύξουμε το δικό μας μοντέλο στον τομέα της υγείας, της παιδείας κτλ. Ό,τι τέλος πάντων είναι σημαντικό για μια κοινωνία. Μεταλλευόμενοι όμως την σα θα πρέπει να κάνουμε ένα πιο βαθύ προβληματισμό ε, και για το μέλλον της αναπτυξής συνεργασίας και εν γέννη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Νίκ Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση ευθυγραμμίζεται με την ανακοίνωση περί κοινωνικής προστασίας στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ενώσης που θετήθηκε πέρσι τον Αύγουστο με συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση αυτού διότι καλύπτει πολλά από τα αναφερθέντα συμπεριλαμβανομένη και της υποστήριξης της τριγωνικής συνεργασίας. Και όπως λέει και η έκθεση, να σας πω ότι DEFCO, στην ΤΕΦΚΟ παριστάμεθα στις συνεδριάσεις ε, του φορέα που αφορά τη συνεργασία. Το Φεβρουάριο στη Νέα Υόρκη έγινε συνεδρία, συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα, αφορά τη διοργανική συνεργασία. Συγκεράζει όλους τους φορείς της αναπτυξιακής συνεργασίας, τους διεθνείς φορείς, ενοποιημένα και συζητούν το θέμα προς ενημέρωσή σας. Τούτου λεχθέντος. Κάποια σχόλια που ίσως να σας βοηθούν, ελπίζω. Πρώτον, ένα τα σημαντικότερα. Πώς είναι βασικό θέμα η κοινωνική προστασία ε, στις συζητήσεις τις μελλοντικές Η συζήτηση περί ανισοτήτων, που είναι και γραμμή προβληματισμού, όπως είδαμε και στη συνάντηση του περασμένου μήνα στην Κοπενχάγη, η ανισότητα και συζήτηση αφορά την κοινωνική προστασία, λόγω του ρόλου που παίζει στην ενίσχυση της ισότητας και στην ανακατανομή του πλούτου Η κοινωνική προστασία στην αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να εξεταστεί. Είναι περίπλοκο το ιστορικό. Σε πολλέ χώρε Αφρική, οι έννοιε κοινωνική προστασία, όπω βλέπουν αυτή την ανάπτυξη, λειτουργούσε ω φορέα μείωση τη ένδυα, όπω το βλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα. Δίκτυα ασφαλεία. Άλλοι αναπτυξιακοί φορεί λένε κοινωνική προστασία και σχετικά προγράμματα. Δεν χρησιμοποιεί το δίκτυο ασφαλεία. Προγράμματα τριετή ή με περισσότερη διάρκεια έχουν στόχο συγκεκριμένε μερίδε του πληθυσμού και θέλουν να βγάλουν αυτά τα τμήματα του πληθυσμού από την ένδυα ανάλογα με τον ορισμό τη ένδυα. Κλασικό παράδειγμα. Σε μεγάλη κλίμακα. Αιθιοπία. Με τα προγράμματα τα παραγωγικών δικτύων ασφαλείας που στηρίζουμε χρηματοδοτείται 100% από τους Αφορά 8 εκατομμύρια ανθρώπους και τους προστατεύει από την ασυτεία και την πείνα. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, όπως διερωτώνται στην Αιθιοπία και διερωτώμεθα κι εμείς. Γιατί η κοινωνική προστασία αφορά την προστασία κατά των κλειδονισμών κατά τη διάρκεια της ζωής. Περί αυτού πρόκειται. Άρα δεν αφορά μόνο τη μείωση της ένδυας. Πρέπει να κινηθούμε και στην προστασία κατά ευαλωτότητας, κλονισμών κλπ για τη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί είναι κρίσιμο. Διότι ακούγονται κάποιες επικρίσεις. Πώς μετράτε η ένδυα σε εθνικό επίπεδο. καλύπτει αυτούς που είναι μόλις πάνω από τη γραμμή της ένδυα, όπως είπε και ο Σκοβαλιών, υπεύθυνο τη Παγκόσμια Τράπεζας. Αυτοί που είναι στα όρια, είναι ευάλωτοι. Αυτό πώς εξετάζεται. Διακοιμάσει κατά τη διάρκεια της ζωής. Ας πούμε, αν κάποιος οραστεί σοβαρά στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων που είναι στα όρια, θα πέσουν αυτοί οι άνθρωποι στη φτώχεια. Και αυτό πρέπει να το καλύπτουμε. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ χωρών με μικρό εισόδημα και άλλων με μεσαίο εισόδημα. Διότι πολλέ χώρε ε, και κυρίω Αφρική ανεβαίνουν προ το μεσαίο εισόδημα, όπω είναι η Γκάνα, η Σβάζιλαντ, η Αγγόλα είναι στο μεσαίο επίπεδο εισοδήματο, ε, σύμφωνα με την Αφρικανική Τράπεζα ε, Ανάπτυξη. Και εκεί είναι τεράστιο το θέμα χρηματοδοτήσεω κυρίω από τον ιδιωτικό τομέα και από τι αποταμίευσει. Διότι υποστηρίζουμε κυρίω χώρε με χαμηλό εισόδημα. Για υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία. Στι χώρες καλύπτονται από του δωρητέ. Αυτά στι χώρε με χαμηλό εισόδημα. Αν περιπλακεί τώρα η κάλυψη λόγω του ότι η χώρα ανέβηκε σε μέσο επίπεδο, πρέπει να εξεταστεί και πώ γίνεται η χρηματοδότηση. Γιατί εκεί χρηματοδοτούνται κυρίω από ποταμιεύσει κλπ. Στι χώρε μεσαίου εισοδήματο πρέπει να δούμε τι γίνεται. Κίνα, Φερρυπίν. Την υποστηρίζουμε ακόμα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν το σύστημα κοινωνική προστασία γιατί ξέρουν ποια προβλήματα εμπεριέχονται. Όταν κινούνται προ αυτό το μέσο εισόδημα οι χώρε εμείς τους αφήνουμε εκτός διμερούς ενίσχυσης, διότι δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο πλαίσιο του προγράμματος για την αλλαγή. Εξακολουθούν να είναι χώρες παρόλο που είναι στο επίπεδο μέσου εισοδήματος, όπου υπάρχουν όμως πολύ ψηλά ποσοστά ένδυας. Και άλλα δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, η κοινωνική, το κοινωνικό συμβόλαιο που αναφέρθηκε. Κάτι πολύ θετικό συμβαίνει στην Αφρική. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις θέλουν να αλλάξουν. Από μικρά σχήματα κοινωνικής προστασίας που βοηθούν να βγουν οι άνθρωποι από την ένδια θέλουν να βγουν σε εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας. Τώρα αν θέτουν όρια, ε, κατώτατα όρια ή όχι. Θέλουμε να, συστη... να τις υποστηρίξουμε ούτως ή άλλως. 23 Φεβρουαρίου παρουσιάσαμε μελέτη σχετικά με την κοινωνική προστασία στην υποσαχάρη Αφρική. Σε μια συνεδρία στην Αντίσα Μπέμπα παρουσιάσαμε την έκθεση. Καλέσαμε λίγες κυβερνήσεις. Αυτές με τις οποίες συνεργαστήκαμε. Αλλά ήρθαν και αυτοπρόσκλητοι α, πρωθυπουργοί και υπουργοί. Είχαμε δει τρεις από αυτούς. Τεράστιο ενδιαφέρον. Οι χώρε θέλουν μεγαλύτερη ισότητα, αλλάζει το περιβάλλον. Θέλουν να αντιμετωπιστούν και βασικά προβλήματα. Και αυτό μέσω κοινωνική προστασία. Θεωρούν ότι έχει και πολιτική αξία. Κερδίζουν ψηφοφόρου. Το είπε ο Υπουργό τη Γκάνα, μάλιστα. Η κοινωνική προστασία, μα είπε, είναι στην εκλογική μα πλατφόρμα. Και γι' αυτό κέρδισε και ο Πρόεδρο, μα είπε. Ενδιαφέρον. Μα είπε η κυρία, μάλλον. Έχουμε σταθερότητα και είμαστε καλύτερα. Είμαστε στο μέσο εισόδημα και μπορούμε να τα αντέξουμε οικονομικά. Ενδιαφέρον το σχόλιο της Υπουργού. Γιατί τα λέω αυτά. Α, και κάτι άλλο να σας ενημερώσω. Και διάφορα όσον αφορά την κοινωνική προστασία και τα διάφορα κενά που υπάρχουν και τα όρια κοινωνικής προστασίας, τα εθνικά. Μια σύσταση θετήθηκε ομόφωνα στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας πέρσι Πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στην εμπειρογνώμονα στην κυρία Μπαστάλη, για να μας ε, πει κάποια πράγματα ακόμα. Για 5-6, για 7 λεπτά μάλλον. Για το κομμάτι για τον ειδικό τομέα, Κοινοβούλιο μου ζήτησε να δούμε ακριβώς το θέμα της συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αν διαβάσετε την ε, μελέτη αυτή θα δείτε ότι υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για την ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ε, θεωρητικά υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για το γιατί κάποιος θα ήθελε να παρέμβει ο ιδιωτικός τομέας σε διάφορους βαθμούς ή σε διάφορες, με διάφορες ε, δυνατότητες ε, και το κεφάλαιο αυτό λέει ότι ακριβώς υπάρχει α, ε, ρόλος να παίξει η κυβέρνηση και είναι σημαντικό για, για κάποιους τομείς να διατηρήσει τον έλεγχό τους η κυβέρνηση. Ας πούμε για μη κερδοσκοπικούς ε, μιλάμε για τη συμμετοχή μη κερδοσκοπικών ε, ιδιωτικών οργανισμών, ε, αλλά όταν η κυβέρνηση μπορεί από μόνη της με βοήθεια των δωρητών να, να στηρίξει την κοινωνική ασφάλιση, θα πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο σε αυτέ τι δραστηριότητε. Θα πρέπει να μπορεί να εποπτεύει όλη αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει ότι αυτέ οι παροχέ δίδονται και είναι και μια αλφαπιότητα. Μετά, η ενημέρωση επικεντρώνεται στο τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν ε, τα κυβερνητικά έσοδα. Για το πώς δηλαδή χρηματοδοτούνται τα προγράμματα αυτά από το κράτος. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια έκθεση. Τι μπορεί δηλαδή η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει για να εξασφαλίσει ότι τα κρατικά έσοδα θα αυξηθούν και ότι θα δαπανηθούν σε τέτοιου είδου πολιτικέ. Γιατί βλέπουμε ε, χώρε μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματο να έχουν εισοδήματα, αλλά να μην τα δαπανούν για αυτού του τομεί. Για κοινωνική ασφάλιση, α πούμε, τα έσοδα πάνε αλλού. Ή έχουμε χώρε πολύ χαμηλού εισοδήματο που, που δεν έχουν έσοδα, οπότε πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να τι ενισχύσουμε, να τι βοηθήσουμε να αυξήσουν τα έσοδά του. Υπάρχει μια πληροφόρηση ω προ αυτό και αυτό ακριβώ καταγράφω και στον, στον πίνακα. Βεβαίω όλα αυτά είναι λίγο φλού, γιατί ε, έπρεπε σε μια έκθεση 20 σελίδων να καλύψω όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω το κάθε θέμα θα έπρεπε να τύχει δική του ξεχωριστή ε, έκθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Οπότε θα είναι δύσκολο να είμαι και αντικειμενική, να δώσω πλήρε πληροφορίε, να παραθέσω όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Αλλά ε, συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι πρέπει όντω να υπάρξει περισσότερη δουλειά σχετικά με το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τα έσοδα τα κρατικά και ανέφερα και κάποιες από τις, κάποιους από τους τρόπους ε, και αποκινούμε το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδα κάποιων χωρών μέσω ε, ενίσχυσης των ε, διοικητικών δομών, των ενίσχυσης των φορολογικών συστημάτων τους κτλ. Και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Τώρα, σχετικά με τον ορισμό της κοινωνική προστασίας, βεβαίως υπάρχει μια έτσι, ιδεολογική πτυχή σε όλο αυτό. Έχουμε δει μια εξέλιξη στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξης από οργανισμούς που κυρίως επικεντρώνονται στη διαχείριση κινδύνου και μιλούν ελάχιστα για την κοινωνική προστασία. Αυτοί έχουν αρχίσει και προχωρούν προς μια πιο ένα πιο ευρύ ορισμό της κοινωνικής προστασίας και της πρόθεσής της. Οπότε βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή. Η κρίση η ίδια νομίζω ότι έχει δείξει ότι μπορεί τα πράγματα να κινηθούν είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Σε κάποιες περιπτώσεις αποτέλεσαν ε, τον κινητήρο μοχλό για την ενίσχυση των κοινωνικών συστημάτων στις χώρες με χαμηλό εισίδημα, για παράδειγμα. Και αυτή η κρίση που περνούμε, είδαμε ότι σε κάποιες ε, χώρες βοήθησε να γίνει αυτό ακριβώς. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η κρίση αυτή για να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων είναι ακριβώς αυτός. Να, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση έτσι ώστε να προωθήσουμε μια πιο δίκαιη, καθολική, ισότιμη ε, κοινωνική προστασία και να έχουμε βεβαίω και ένα ε, δίκτυο ασφαλείας για όλους. Σε σχέση τώρα με, τον, ε, με την χρηματοδότηση από και γενικά για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, ε, αναφέρεται και στην έκθεση αυτό, η χρηματοδότηση από ήταν ζωτική σημασίας... για να ξεκινήσουν τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας δεν μπορώ να τα ονομάσω πολιτικές, ήταν κυρίω project ή προγράμματα. Αυτό που δεν ήταν τόσο επιτυχέ ήταν η μετάβαση των προγραμμάτων σε εθνικές πολιτικές, η μετάφρασή τους σε εθνικές πολιτικές και η ε, εθνική ε, ιδιοκτησία αυτών των προγραμμάτων. Δηλαδή, οι, πρέπει να μπουν σε εταιρική σχέση με τις κυβερνήσει. Να παίξουν δηλαδή το ρόλο του κινητήριου μοχλού για να ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα, αλλά με, μια, με ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο όραμα το οποίο έλειπε παλαιότερα από τα προγράμματα. Οι δωρητέ μέχρι τώρα ήταν υπέρ προγραμμάτων που είχαν άμεση, άμεση συνέπεια στην αντιμετώπιση της φτώχεια, βραχυπρόθεσμη δηλαδή. Αλλά αν δούμε τον αρχικό στόχο του τι είναι η κοινωνική πολιτική και τι είναι η κοινωνική ασφάλιση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια προοπτική μέσο μακροπρόθεσμη. Και αυτό μπορεί να γίνει υιοθετώντα ένα πιο μακροπροθεσμό όραμα, δρώντας από κοινού με τις, ε, με τις κυβερνήσεις και συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις εταιρικές σχέσεις, αυτές τις συμπράξεις, ένα σχέδιο μετάβασης, μετάφρασης αυτών των προγραμμάτων σε προγράμματα ή πολιτικές εθνικές. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και βεβαίως σχετίζεται και με την συζήτηση για την ε, κυβερνητική, για την κρατική χρηματοδότηση, καθώς επίσης και την αύξηση των εσόδων των χωρών για την παροχή κονδυλίων στην κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στο σημείο 11 τη συνεδρίασή μα, τη ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γενική Συγήτρια για τον προπολογισμό, την κυρία Αν Γένσεν, που την υποδέχομαι θερμά. Φέτος η συζήτηση επί του προϋπολογισμού θα είναι δύσκολη διότι είμαστε στην αβεβαιότητα. Όπως το πολιετές πλαίσιο δεν έχει εγκριθεί ακόμα, αλλά βασίζομαι στην κυρία Γένσεν, η οποία θα μας διαφωτίσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με αφήσατε να έρθω εδώ και να συζητήσουμε σύντομα τον προϋπολογισμό. Πράγματι, ο προϋπολογισμός του 2014 πράγματι είναι αβέβαιος, εφόσον δεν έχουμε το πολιετές πλαίσιο, δεν έχουμε την ομοθεσία, δεν έχουμε τίποτα άρα πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε το ψήφισμα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, απορρίψαμε τα προτινόμενα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ψηφίσαμε κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό του 2014 ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει για τον ελόγο προπολογισμό 2014 ένα προϋπολογισμό που θα βασίζεται στην πρότασή τη για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι αυτό έχουμε επιτάπητος τώρα και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ανησυχεί τα μάλα διότι δεν μπορούμε να δειχθούμε έτσι ε, αψήφιστα τα όσα προήλθαν από τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο δικό σας τομέα συγκεκριμένα, κατηγορία 4 του προϋπολογισμού, βλέποντας τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν μόλις 3% η αύξηση μέχρι το 2020 εν συγκρίση με αυτή την προγραμματική περίοδο άρα πολύ μικρή αύξηση σε έναν τομέα όπου επανειλημμένα έχουμε διαπιστώσει ότι τα πάντα ήταν στενά και θα έχουμε σίγουρα κάποια έλλειψη ευελιξίας διότι το απόθεμα ανάγκης μπήκε στην κατηγορία αυτή. Άρα πολλά πρέπει να εξεταστούν όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι κάτι που θα επηρεάσει και τον προϋπολογισμό του 2014. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωρίζω ότι ήταν μια πρόταση που δεν έγινε πρόσδεκτη σε αυτή την Επιτροπή. Θεωρήθηκε άκρος μετριοπαθής Μιλώντας με επιτρόπους τώρα σχετικά με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μου τόνισαν οι επίτροποι ότι χρειαζόμαστε χρήματα για ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να βρούμε μια λύση για το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να ενισχύσουμε κάποιους τομείς που είναι αγαπητοί σε αυτή την Επιτροπή, αλλά είπαν ότι κάποια προγράμματα γειτονία δεν εφαρμόζονται και τόσο καλά. Πολύ συχνά όταν δίνουμε τα χρήματα και δίνουμε τα κονδύλια, εμπεριέχεται ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτά τα προγράμματα, αλλά μου είπαν ότι τα προγράμματα σου μην εφαρμοζόνται σωστά, θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον ε, προπολογισμό του επόμενου έτου, Αύριο θα διεξαχθεί ο πρώτο τρίλογος που θα είναι πολύ γενικό το πλαίσιο των συζητήσεων. Θα δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση, πώ θα κινηθούμε εντό του προπολογισμού. Είναι σαν το Συμβούλιο να μην ανακάλυψε ότι υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνα. Βασικά τα πάντα τα αντιμετωπίζουν όπω τον παλιό καιρό. Το Συμβούλιο ότι έχει το λόγο για την αγροτική πολιτική και εμεί έχουμε το τελευταίο λόγο στα άλλα. Ενώ η συνθήκη τη Λισαβόνα το πνεύμα της συνθήκης της Αβώνας πραγματικά ποιο είναι ότι ξεκινάμε σοβαρή συζήτηση για κάθε γραμμή του προπολογισμού. Είμαστε δύο φορείς ισότιμοι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Πρέπει να πω όμως ότι από τότε που ετέθησε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας δύο από τις τρεις φορές δεν είχαμε προπολογισμό για τον επόμενο χρόνο και είναι ανόητο πραγματικά. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν πάρα πολύ κοντά από την αρχή. Δεν φαινόταν να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι γελία η αντιμετώπιση από πλευρά Συμβουλίου. Δεν θέλει να ξεκινά τις διαπραγματεύσεις παρά σε ένα πολύ ε, μεταγενέστερο στάδιο και δεν θέλει να μπει στην ουσία το Συμβούλιο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και τη βοήθεια των ε, ειδικών επιτροπών πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι σαν κοινοβούλιο για λεπτομερέστερες, πολύ λεπτομερέστερες ε, συζητήσεις. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια που είχα να πω και θέλω να ακούσω τα όσα έχει να πει η Επιτροπή σας και ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για τον προπολογισμό 2014, τον κύριο Λάστρα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γένσεν. Είμαστε ε, ουσιαστικά στην απαρχή της συζήτησης. Θα σας αναφέρω τέσσερις βασικές ιδέες. Πρώτη, είναι ανάγκη και για την αναπτυξιακή συνεργασία και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Έχουμε τα στοιχεία, έχουμε τους αναπτυξιακούς τόσους της χιλιετίας, ε, Έχουμε όλο και περισσότερες ανθρωπιστικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια και είναι προφανείς λόγοι γι' αυτό. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Είπαμε γι' αυτό 0,7 του ΑΕΠΑ για τη βοήθεια. Και αυτός ο νοστός πρέπει να τηρηθεί. Και το Ευρωβαρόμετρο το Οκτωβρίου του 2012 επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες, η δημόσια κοινή γνώμη, στηρίζει, στηρίζει στεναρά την αναπτυξιακή βοήθεια. Και πολλοί ε, θα ήταν υπέρ του να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Άλλη ιδέα που είναι σημαντικό να αντιλάβουμε υπόψη μας. Η αναπτυξιακή βοήθεια, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι επιτακτική ανάγκη και από ηθικής πλευράς. Αν δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα κατά πολλών προβλημάτων, μετανάστευση, φτώχεια, ε, αποξένωση, υποβάθμιση βιωτικού επίπεδου, πρέπει να προστατεύσουμε την αναπτυξιακή συνεργασία. Γιατί ξέρουμε ότι επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι κατά την άποψή μου η αναπτυξιακή συνεργασία και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αποτελεσματικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να το πούμε. Είμαστε αποτελεσματικοί. Μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, είμαστε όμω αποτελεσματικοί. Άρα πρέπει να υπάρξει συνέχεια και νέα δέσμευση. Αυτό το δείξαμε όλες τις πολιτικές ομάδες ε, που εκπροσωπούμαστε εδώ σε αυτή την Επιτροπή και με την ανθρωπιστική συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδίως για το 2014. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τον Ρικάρντο για τα σχόλια. Συμφωνούμε. Όλες οι πολιτικές ομάδες Επιτροπής. Όλοι είμαστε σε επαφή με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και μέσω ημών, κυρία Πρόεδρε, και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Γένσεν για το πώ πλαισιώνεται ο προπολογισμό. Το Συμβούλιο κινείται σαν να μην κατάλαβε ότι υφίσταται συνθήκε Λισαβόνα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το καταλάβουν. σω να μην βολεύει αυτό την Ιρλανδική Προεδρία, για πολλού λόγου, αλλά σίγουρα στην ομάδα μου και σε άλλες ομάδες είμαι βέβαιος υπάρχει το συνέστημα ότι πρέπει να δείξουμε ότι δεν θα επικυρώσουμε τυπικά αυτό που αποφασίζουν αυτοί. Ποιο είναι ένα από τα προβλήματα δεν θα έχουμε περιθώρια στον προπολογισμό που θεωρούσαμε ότι θα έχουμε. Αλλά, εν συγκρίση με αυτό, κανείς σε αυτή την Επιτροπή δεν απευθύνει έκκληση για την εκλογική περιφέρεια. Δεν πρόκειται περί ψηφοθυρίας και ιδίου συμφέροντος. Κάθε μέρα πεθαίνουν 23.000 παιδιά και έχουμε υποχρεώσεις για αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ δεν ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας. Και αν δεν καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να το κάνουμε για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν θα προχωρήσουμε καθόλου προς στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα πολεμήσουμε όλοι μαζί, συλλογικά, όλες οι πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή για να παραμείνει και να αποκατασταθεί ο προπολογισμό και ο πρόεδρος Σούλτς ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για το θέμα. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή ίσω να είναι σε θέση να μας βοηθήσει να σημειώσουμε τέρμα στον αγώνα. Πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει η συνθήκη της Λισαβόνας και δεν πρόκειται να επικυρώσουμε τυπικά τον προπολογισμό. Θέλουμε να επαναξεταστούν τα ανθρωπιστικά θέματα. Δεν είναι κάτι σαν διευθυντικά ταμεία την κοινή αγροτική πολιτική που αφορά τους εκλογείς μας. Αυτό είναι διαφορετικό. Πρόκειται περί ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν πρόκειται περί ιδίου συμφέροντος ούτε περί ε, συλλογής ψήφων. Κύριε Μαρτίνες. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρία σχόλια μόνο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο φίλος Μωρικάρτο και ο κύριος Γκέι Μίτσελ. Πρώτα απ' όλα, στο κοινοβούλιο αυτό κάποιες φορές δεν γνωριζόμαστε όλοι οι συνάδελφοι. Γνωρίζουμε αυτού με του οποίου ε, είμαστε μέλη στην ίδια επιτροπή. Είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με την κυρία Γένσεν για κάποια ζητήματα και η κυρία Γένσεν είναι εγγύηση. Γιατί δεν είναι μόνο άκρο αποτελεσματική και αποφασιστική, αλλά έχει και τη συνείδηση που την ε, παρακινεί ε, να εργαστεί για τα θέματα τα οποία Μα απασχολούν και μας εδώ στην Επιτροπή μας. Εμένα με καθησυχάζει κατά κάποιο τρόπο που η κυρία Γένσεν είναι αυτή που σε αυτές τις τόσο δύσκολε, τόσο ιδιαίτερες συνθήκες χειρίζεται αυτό το τόσο λεπτό θέμα. Δεύτερον, ε, έχω ένα πάρα πολύ απεσιόδοξο προέστημα για το τι γίνεται και για το τι πρόκειται να γίνει. Το Συμβούλιο έκανε μια πρόταση που είναι απαράδεκτη πολύ απλά και είναι και αναξιοπρεπής και αντίθετη με τους ε, κανόνες της συνθήκες και μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανείς αυτή την πρόταση του Συμβουλίου. Και πρέπει να ομολογήσω εδώ, επειδή δεν είμαστε και πολλοί, μπορώ να το ομολογήσω έτσι με πιο μεγάλη ηρεμία, πρέπει να σας ομολογήσω ότι εγώ εμπιστεύομαι ελάχιστα, ε, τέλος πάντων έχω ελάχιστη πίστη στο ότι θα μπορέσει ε, το Κοινοβούλιο να ε, εμείνει σε αυτή τη θέση του. Αυτό που προβλέπω είναι το εξής σενάριο. Το Συμβούλιο θα μας δώσει 4-5 καραμέλες ως δωράκι απλά και μόνο για να πει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου κάτι πήραμε, κάτι καταφέραμε. Ξέρετε, αυτή η τακτική είναι όλο και πιο επικίνδυνη. Και βλέπουμε να παίζεται το ίδιο παιχνίδι σχεδόν σε όλες τις χώρες. Κάνουν μία πρόταση που είναι πονίδιστη, που είναι ντροπή και μετά δίνουν κάτι, κάτι της και λένε «Α, ωραία, κάτι μας δώσανε, ωραία, θα το δεχτούμε». Αυτό το οποίο με ανησυχεί μεταξύ άλλων, είναι ότι μια από απαιτήσει μα που φυσικά και δεν πρόκειται να επαναχωρήσει σε αυτό το Συμβουλίο, είναι το θέμα της ευελιξίας. Και στο θέμα της ευελιξίας, αυτό που μπορούμε να πετύχουμε για αυτό που μας απασχολεί εμάς, δηλαδή για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, θα χάσουμε ε, στην ευελιξία, γιατί είμαστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Δηλαδή, για την ανθρωπιστική βοήθεια και την, ε, και την αναπτυξιακή συνεργασία, ό,τι προβλέπετε θα κοπεί, με, θα ψαλιδιστεί λόγω της ευελιξίας, αν θέλετε. Για θέματα που για άλλους, ε, για τους κυβερνήσεις ή ίσως και φοβούμε για κάποιους βουλευτές εδώ, θεωρούνται περισσότερο προτεραιότητα. Γιατί αυτά που κάνουμε εμεί είναι πιο πολύ για πολίτε που δεν είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απομακρυσμένοι, ζουν σε μακρινέ χώρε. Αυτή είναι η ανησυχία μου και ελπίζω να κάνω λάθο. Εγώ προσωπικά πάντως είμαι απόλυτα δεσμευμένο και νομίζω ότι και πολλοί συντροφοί μου δεν θα χωνέψουμε τις ε, τέσσερις καραμέλες, δεν θα ε, αρκεστούμε σε αυτές. Θέλω να κάνω στην κυρία Γένσεν το εξή ερώτημα. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ψηφίσει τον προπολογισμό, καταλαβαίνω ότι για το 2014 θα λειτουργήσουμε με τον προπολογισμό του 2013. ο οποίος είναι καλύτερος ή τέλο πάντων δεν είναι καλύτερος, δεν ξέρω, θέλω να μου τα πει κυρία Γένσεν τουλάχιστον για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, αναπτυξική συνεργασία, είναι καλύτερο ο προπολογισμό του 2013 από ότι θα ήταν ο αντίστοιχος προπολογισμό του 2014. Εάν αυτός ο προπολογισμό βασιστεί στην προσφορά που μας έχει κάνει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο για την επταετία. Θέλω λοιπόν να μου το διευκρινίσει αυτό η κυρία Γένσεν. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση έχω ένα ακόμη επιχείρημα στα χέρια μου να πω εγώ δεν τον ψηφίζω αυτό τον προϋπολογισμό, αυτή την πρόταση του Συμβουλίου, ούτε και με τι καραμελίσει που θα μου δώσουν. Γιατί για το 2014, αν δεν τον ψηφίσουμε, θα έχουμε το προπολογισμό για την ανάπτυξη που θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που θα έχουμε να ψηφίσουμε τον προπολογισμό για το 2014. Άρα αυτό είναι ένα επιχείρημα ακόμη για να μην ψηφίσει το Κοινοβούλιο αυτό που μας προσφέρει το Συμβούλιο. Αν επαναλαμβάνω με τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν, η διόρθωση που θα μας παράσουν, θα μας προσφέρουν δεν είναι τόσο ευρεία που δεν νομίζω ότι θα είναι ούτως ή άλλως. Έχω λίγες ελπίδες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γένσεν και θέλω να την εμψυχώσω, να τη πω ότι έχει όλη την υποστήριξή μας. Αλλά θέλω να διευκρινίσω το εξή. Εάν δεν ψηφίσει το Κοινοβούλιο τι δημοσιονομικέ προοπτικές 14-20, θα έχουμε περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη και για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2014 συγκεκριμένα. Και βέβαια το ίδιο θα ισχύσει για το 2015 και το 2016. Αν είναι να έχουμε περισσότερους πόρους από αυτού που θα έχουμε, αν ψηφίσουμε, αυτό ε, είναι θετικό να το ξέρουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Μαρτίνες. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Η κυρία Κάθριν Μέτε Πέριγκεν, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο από πέντε λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί τη τριμερή ιδιόλογα από τη Γενική Διεύθυνση για τον Προπολογισμό DG Bodge χειρίζεται τη θέση μας όσον αφορά όλα τα κονδύλια του προπολογισμού και όχι μόνο αυτή που αφορά την εξωτερική βοήθεια και την αναπτυξιακή. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, των απροσμετρήτων για την υλοποίηση του προπολογισμού του 2014, διότι όπως επισημάνεται πολύ σωστά δεν έχουμε κανένα πλαίσιο δημοσιονομικό, εξαιρετική περίσταση στην ιστορία τη θεσμική μας όπως είπε και ο Μπαρός, ο πρόεδρος Μπαρός, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τα πάντα για να παίξει επικοδομητικό ρόλο στην έγκριση του προπολογισμού 2014. Για να έχουμε ένα πλαίσιο να κινηθούμε μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Προσωπικά θα εξέφραζα την ίδια ανησυχία που εξεφράστηκε ελήψη προϋπολογισμού του 2014 θα έχουμε παράταση του εκείνου του 2013 από αυτές τις περιστάσεις θα είναι δίκοπο μαχαίρι. Απαντώντας λοιπόν στην, κυρία Γέντσεν, αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προσέχουμε προς τα που κατευθύνουμε το δίκοπο μαχαίρι. Λοιπόν, ε, στρέφουν όλοι το βλέμμα προς την κυρία Γένσεν για να δώσει απαντήσεις στα τόσο σημαντικά ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που τονίσατε και την ηθική πτυχή αυτής της υπόθεσης. Νομίζω ότι πάντα πρέπει να την ε, θυμόμαστε. Τι θα γίνει αν δεν πούμε ναι αν δεν υπάρξει ε, συμφωνία. Θα μείνουμε στο όριο του 2013. Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει με τις νομοθετικές εκθέσεις, να ε, ολοκληρωθεί η νομοθεσία και να πει ότι θα πρέπει να συνάδει αυτή η νομοθεσία με τα όποια όρια είναι αυτά που έχουν τεθεί. Αν δεν είναι είτε αν δεν έχει αποφασίσει η Κομισιόν για το πολιετές δημοσιονομικό ταμείο ή, για, ή το Συμβούλιο, τότε θα παραμείνουμε στα όρια που έχουν δοθεί για το έτος 2013. Τώρα το Συμβούλιο επιμένει ότι αυτό δεν υπάρχει ως επιλογή. Αν πείτε όχι, θα σταματήσουμε οποιαδήποτε νομοθετική εργασία συχαίνονται το ότι εμείς λέμε «Μα αφού υπάρχει το όριο του 2013 μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό». Πραγματικά συνέχεια μας λένε «Όχι, αυτό δεν γίνεται». Που ουσιαστικά α, μου λέει εμένα ότι τους ανησυχεί. Ε, το ότι μπορεί να πούμε και όχι. Βεβαίως όλοι μας θέλουμε να βρούμε μια λύση, αλλά όχι την οποιαδήποτε λύση. Ε, μπορεί κανεί να πει ότι το όριο του 2013 όντω δίνει περισσότερα κονδύλια. Περίπου 10% παραπάνω. Αλλά είναι διαφορετική η κατανομή. Ε, περισσότερα κονδύλια δίδονται στην ε, Γεωργία και λιγότερα στο Connecting Europe, στην έρευνα κτλ. Για τα δικά σας τα θέματα δεν θα ήταν τεράστια διαφορά. γιατί ούτως ή άλλως δεν σας έχει δοθεί μεγάλη αύξηση, οποιοδήποτε και αν είναι η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι. Και αυτό για μένα σημαίνει ότι καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση. Βεβαίως πρέπει να διαπραγματευτούμε για να βρούμε λύση. Και αυτό γίνεται ακριβώς στις διαπραγματεύσεις για το MFF. Ο κύριος Μπέγκε και ο κύριος Κάλφιν συναντώνται τακτικά οι δύο ε, ε, εισηγητές του Κοινοβουλίου με τους ε, εξειδικευμένους εισηγητές των δύο επιτροπών για να συντονιστούν, για να δουν ποιοι είναι αυτοί οι πέντε ή εφτά τομείς που πρέπει να βρούμε μια κοινή άποψη. Ο δικός σας ο τομέας θα μπορούσε να είναι ένας, που, ένας τομέας που θα μπορούσε ίσως να του δοθεί μια κάποια ευελιξία γιατί διαφέρει η κατάσταση που αντιμετωπίζεται από χρόνο σε χρόνο. Και όταν μιλούμε για ευελιξία, είναι ακριβώ ο δικό σου τομέα που χρειάζεται ευελιξία, γιατί ακριβώ πολλέ φορέ χρησιμοποιεί την ευελιξία του ενό χρόνου ή τα κονδύλια του ενό χρόνου για τον άλλον. Αλλά δεν ξέρει κανεί τι θα γίνει. Κανεί δεν ξέρει πότε μπορεί να να γίνει πόλεμος κάπου που να χρειάζεται μια χώρα περισσότερα κονδύλια, πότε μπορεί να γίνει κάποια να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση. Ανά χρόνο τα πράγματα αλλάζουν, οπότε γι' αυτό χρειάζεστε ευελιξία. Αλλά για τον ετήσιο προπολογισμό είναι δύσκολο όταν δεν υπάρχει ούτε καν γενικό πλαίσιο. Βεβαίω μπορεί κανείς να υποβάλει μια πρόταση και να ξεκινήσει νέα προγράμματα με βάση την νέα νομοθεσία. Εμείς σε όλες τις επιτροπές ε, και τις δική σας συμπεριλαμβανομένες προτείνουμε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την νομοθετική βάση. Γιατί μέχρι 1η Πρώτου 2014 θα πρέπει να έχουν καταλήξει. Ανεξάρτητα από το ποιο πλαίσιο τελικά θα υπάρξει το οικονομικά. Νομοθετικά θα πρέπει να έχει γίνει αυτή η δουλειά. Γι' αυτό έχετε την, τη δύναμη, το Κοινοβούλιο έχει τη δύναμη ακριβώς να δράσει στο, στο πεδίο της νομοθετικής εργασίας και πρέπει να συντονιστούμε σωστά έτσι ώστε να έχουμε καλή, σωστή νομοθετική βάση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Merci. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες και όλους. Διακόπτουμε τη συνεδρίασή μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9 θα υπάρξει μια κοινή ακρόαση. Ντεβε και Κρίμ. Θέμα διαφθορά και το ξέπημα βρώμικου χρήματος, εγκληματικότητα. Θα υπάρξουν προσωπικότητα, προσωπικότητες επιφανείς που θα έρθουν να μας μιλήσουν. Αύριο το πρωί τα λέμε σε αυτή την αίθουσα, 9 η ώρα. Καλό βράδυ.